Καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την απόψηνή μας συνεδρίαση. So, ladies Κυρίες και κύριοι, καλό ε, απόγευμα. Σας χαιρετίζω όλους και σας καλωσορίζω. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να καλωσορίσω την οριστή εκπρόσωπο κυρία Γκάμπριελ ο φάκελος δε που της έχει προταθεί από την πρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λάιεν, είναι η καινοτομία και νεολαία. Θα ήθελα επίσης να καλώσω την κυρία Φερχάνα, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, καθώς επίσης και τα μέλη της ε, ίδιας Επιτροπής. Και πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε κοινή ακρόαση με τις ε, δύο επιτροπές σήμερα το βράδυ. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους, ε, καθώς ε, επίσης καλωσορίζω και όλους όσοι παρακολουθούν τούτη την ακρόαση, είτε ε, διαζώσεις είτε μέσω του διαδικτύου. Εμείς είμαστε ε, οι υπεύθυνε επιτροπές ε, για αυτήν την ακρόαση, καθότι είμαι θα υπεύθυνη για θέματα πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έρευνα και την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζομαι ότι αυτό το τρίγωνο της γνώσης, της εκπαίδευσης και της έρευνας και της καινοτομίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικός είναι και ο νέος ψηφιακός ε, κόσμος, ε, ε, θέματα τα οποία έχει προωθήσει ιδιαίτερα η πρόεδρος κυρία Φόντερ Λάγεν στο θεματολόγιο της. Έχουμε, θα αξιολογήσουμε τις κεντρικές γραμμές της πολιτικής της Κομισιόν, καθώς επίσης και την σε πρόσωπο όσον αφορά τρία στοιχεία. Επίσης θα αξιολογήσουμε την γνώση της όσον αφορά τους φακέλους της καθώς επίσης και ε, τις επικοινωνιακές της ικανότητες. Ε, να υπενθυμίσω ότι ε, έχει ήδη απαντήσει γραπτά σε ένα πρώτο ερωτηματολόγιο οριστής εκπρόσωπος και αυτό έχει μοιραστεί σε όλες τις γλώσσες και, γλώσσες και επίσης η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει ασκήσει οποιαδήποτε αναστολή όσον αφορά την ε, ακρόαση αυτή. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Γκάμπριελ για 15 λεπτά. Βεβαίως ε, θα υπάρχουν και άλλα 5 λεπτά στο τέλος της συνεδρίασης. Μετά από την εισαγωγή που θα κάνει η κυρία Γκάμπριελ θα έχουμε 25 ερωτήσεις από τα μέλη των δύο επιτροπών κάθε μέλος ή μάλλον κάθε ερώτηση ε, θα έχει πέντε λεπτά, μία ερώτηση, με ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο για την ε, απάντηση και μετά επίσης μία συμπληρωματική ερώτηση ενός λεπτού με απάντηση συμπληρωματική ενός λεπτού. Ε, ξέρω ότι και εγώ η ίδια αλλά και η κυρία Φερχάγεν είμαστε, ε, είμαστε αποφασισμένες να τηρήσουμε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και οπωσδήποτε πρέπει όλοι να τους σεβαστούμε τους κανόνες αυτού. Θα έχουμε λοιπόν ένα πρώτο γύρο 7 ερωτήσεων από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων μέσω των συντονιστών, επίσης των δύο επιτροπών και μετά 18 ερωτήσεις, ένα δεύτερο γύρο ε, που θα αφορούν όλες τις πολιτικές ομάδες καθώς επίσης και εκπροσώπους των μη εγγεγραμμένων. Έχουμε διερμηνία σε 23 ε, γλώσσες και επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σας. Επίσης μην λυμσμονείτε ότι προβλέπετε διερμηνία, ότι αυτά που θα πείτε θα πρέπει να περάσουν από την διερμηνία και, από τους διερμηνείς και επομένως παρακαλώ να μην μιλάτε με υπερβολική ταχύτητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Σαμπίνα Φερχάνα έτσι ώστε να κάνει και εκείνη τις εισαγωγικές της παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, σαφή ε, διευκρίνηση του πώς θα λάβει η χώρα η ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ εξ της Επιτροπής Πολιτισμού την υποψήφια Επιτροπό, την κυρία Γκάμπριελ και ξέρετε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τα θέματα καινοτομία νεολαία και αθλητισμού, άρα είστε πάρα πολύ κεντρικοί για τα δικά μας θέματα της δικής μας Επιτροπής. Και Δυστυχώ, θέλω να κάνω μια προσωπική παρατήρηση, ο πολιτισμό ε, και η εκπαίδευση και η έρευνα δεν έχουν ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο. Ε, και γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου σας και παρά το γεγονός ε, ότι κυρίως έχουμε θέματα νεολαίας, Αυτά φυσικά αφορούν όλους τις πληθυσμιακές ομάδες και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τα τονίσω αυτό. Έχουμε πολλές προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες. Θα αναπτύξουμε έναν κοινό εκπαιδευτικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επεκτείνουμε τα πολιτισμικά προγράμματα και επίσης θέλουμε να επεκτείνουμε το, την πολιτισμική μας κληρονομιά θα στον τομέα του αθλητισμού θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πιο πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στους νέους και να πραγματοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις γραπτές σας απαντήσεις, τις ερωτήσεις τις οποίες σας θέσαμε ε, πριν από την σημερινή ακρόαση και τις επόμενες τρεις ώρες ελπίζω να ακούσουμε πιο πολλές ε, θέση σας για τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Ήτρε. Και χαίρομαι που η ακρόαση αυτή θα απαντήσει, ελπίζουμε, τι βασικέ μα ερωτήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να θυμίσω την κυρία Βάλεαν και εγώ. Θα τηρήσουμε πολύ αυστηρά τα χρονικά πλαίσια, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Sabine. So... Uh, Ευχαριστώ πολύ, Σαμπίνε. Κυρία Γκάμπριελ, θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλιάν, κυρία Πρόεδρε, κυρία Βερχάιεν, κυρίες και κύριοι, συντονιστές και μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας και Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, Καθοδόν προς εδώ, θυμήθηκα που ακολουθούσα τον ίδιο δρόμο στις 20 Ιουνίου του 2017 και διεξήγε τότε ακρόασή μου όταν ήμουν υποψήφια επίτροπος. Αυτά τα δύο χρόνια και τρεις μήνες συνεργαστήκαμε σε πνεύμα συνεργασίας, συμβιβασμού και κοινού οράματος για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους με τους οποίους συνεργάστηκα σε πολλά θέματα ψηφιακά. Ήταν μέρες που περάσαμε και νύχτες περάσαμε μαζί, αλλά πολύ συχνά άξιζε τον κόπο η όλη προσπάθεια. Ήταν καρποφόρες οι συζητήσεις με πολλούς από εσά και ελπίζω αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί. Και το εύχομαι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Βουλγαρίας και τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μπερίσοφ που με να είμαι υποψήφια επίτροπο από τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ την, Ursula, την κυρία Βοντερ Λάιεν, την υποψήφια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συνάθρισε τη γενοτομία και την έρευνα μαζί με την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την νεολαία, τα θέματα που αφορούν την νεολαία. Και που μου ανέθεσε αυτό το πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο. Δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησα με την ψηφιακή ενία αγορά Χαίρομαι που πολλές πρωτοβουλίες από το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο μπορούν να αποκτήσουν τώρα μια νέα διάσταση και πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες στο διάλογό μας θα εντοπίσουμε νέες ιδέες, εργαλεία, μέσα για τους ερευνητές μας, για τους καινοτόμους μας φορείς, τα πανεπιστήμια, τους καθηγητές, τους δάσκαλους, τους αθλητές, τους νέους, τους καλλιτέχνες και βασίζομαι σε εσά για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κοινό στόχο να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο επιστημών, παιδείας, καινοτομίας, πολιτισμού, αθλητισμού, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων, των πολιτών μας. Σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να ακολουθήσω πάντα τη δική μου προσέγγιση, δηλαδή στο επίκεντρο των πολιτικών πάντα είναι ο άνθρωπος. Δεν θα κάνουμε διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω ούτε οι νέοι ούτε πιο ηλικιμένοι. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η τιμή μου και, ε, που μου κάνετε και με μεγάλη ταπεινοφροσύνη στέκομαι σήμερα μπροστά σας ως υποψήφια επίτροπος ε, υπεύθυνη για την έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την νεολαία και τον αθλητισμό. Πρόκειται να ξεκινήσουμε λοιπόν μια νέα εταιρική ε, σχέση που ευελπιστώ ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο, ε, ε, και ακόμα πιο διαρκής από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό που θέλω θα είναι να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα την, στη συνέχεια της δέσμευσης που είχαμε αναλάβει ήδη στην προηγούμενη ακρόαση. Θέλω να δουλέψουμε για μια Ευρώπη πιο συμπεριληπτική που δεν θα αφήσει πίσω κανέναν ούτε πιο μεγάλο ούτε πιο μικρό. Το φάκελο ε, που μου εμπιστεύτηκε η κυρία Πρόεδρος Βόντερ Λάγεν ε, είναι στην ουσία ένας φάκελος καινοτόμος. Ξεκινάει από τη βασική έρευνα και ε, με την ακτινοβολία των πολιτισμών μας και φτάνει μέχρι την προώθηση της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Συμπεριλαμβάνει προγράμματα πολύ γνωστά όπως το Horizon Erasmus, Creative Europe, Discover EU. Πρόκειται για ένα ε, σύνολο ε, συνεκτικό, το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να προωθήσουμε μέσω της δημιουργίας συνεργειών. Ο κοινό παρονομαστής ανάμεσα σε όλους αυτούς τους τομείς και που αγγίζει σε όλους ε, τους πολίτες της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτή η Ευρώπη των ταλέντων και είναι αυτή η Ευρώπη της καρδιάς. Η Ευρώπη των ταλέντων, γιατί για πρώτη φορά οι πολιτικές του τριγώνου των γνώσεων, εκπαίδευση, έρευνα, έρευνα, καινοτομία βρίσκονται στο ίδιο, στον ίδιο φάκελο. Είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες ε, για την βιωσιμότητα ε, και για την ανάπτυξη. Είναι αυτές επίσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετάβαση στο οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Είναι αυτή αυτές ε, οι μεταβάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του κλίματος και των τεχνολογικών και δημογραφικών εξελίξεων. Αυτά τα ταλέντα τα γνωρίζετε ήδη, είναι οι καθηγητές μας, ε, είναι οι φοιτητές μας, ε, είναι οι καινοτόμοι, αυτοί που ασχολούνται με την καινοτομία, είναι οι ερευνητές μας. Αυτή η Ευρώπη των ταλέντων λοιπόν εψυχώνει την ε, νεολαία μας, τους δημιουργούς μας, καθώς επίσης και τους καλλιτέχνες, όπως και τους αθλητές μας, όποιο αθλητικό επίπεδο και αν έχουν αυτοί. θα ήθελα ε, ήδη τώρα να σας πω εν συντομία ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις κατά την άποψή μας. Πρώτα απ' όλα ε, η διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ε, στην ηγεσία του κόσμου. Εμείς είμαστε μονάχα το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά 20% της έρευνας και της ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς επίσης και ένα τρίτο των επιστημονικών δημοσιεύσεων αφορά την Ευρώπη. Πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες και την Κίνα που όμως μας πλησιάζουν με πολύ γοργό ρυθμό. Είναι θεμελιώδου σημασία η Ευρώπη να διατηρήσει αυτή την ηγετική της θέση γιατί βεβαίως από την έρευνα ε, προέρχεται και η ε, γνώση. Το δεύτερο, η δεύτερη πρόκληση είναι ε, και παράδοξη. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτήν την θέση μας θα πρέπει οπωσδήποτε το ε, ερευνητικό μας πρόγραμμα να παραμείνει όσο γίνεται πιο ανοιχτό και σε σχέση με σήμερα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις καινοτόμες επιχειρήσεις μας. Η Ευρώπη βρήθη νέων ε, επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών που θέλουν να αναπτυχθούν. Ε, πρόκειται όμως για επιχειρήσεις οι οποίες πολλές φορές αναγκάζονται ε, να απομακρυνθούν λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τους μισθούς κλπ. Οπωσδήποτε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ε, για τις νεοφυείς μας επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματίες, για τους ερευνητές μας. Ε, ε, η τρίτη πρόκληση είναι ακριβώς αυτή η διεύρυνση, το widening, να γίνει και μοίρασμα, να γίνει παρτάζ. Στη, η ρήξη, το ρήγμα αυτό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην έρευνα και την καινοτομία είναι μια πραγματικότητα. Εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, η διαρροή εγκεφάλων, οι χαμηλές αμοιβέ αποτελούν μεγάλο πρόβλημα πρόβλημα. δεν είναι εύκολε οι λύσεις. Ε, Στι ε, ημέρες έρευνα και καινοτομία. Ε, εγώ εμπνεύστηκα από αυτά που μου είπαν διάφοροι ερευνητέ σε προγράμματα εταιρικών σχέσεων, προγράμματα teaming καθώς και σε προγράμματα αδελφοποιήσεων. Τους άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατάλαβα ότι η δυναμική τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το η τέταρτη πρόκληση είναι η εμπλοκή των πολιτών και των περιφερειών. Δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή χωρίς ε, να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ότι πραγματικά υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στους κοινούς τους στόχους. Φυσικά αυτό αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή. Γι' αυτό θα ήθελα και σας παρακαλώ, σας προσκαλώ ε, να ακολουθήσουμε μαζί αυτήν την πορεία. Η πέμπτη πρόκληση εγγράφεται στην ίδια λογική ε, και αφορά, σχετίζεται μάλλον με τον γεωπολιτικό ρόλο ε, που έχει κατά νου η κυρία Φόντερ Λάγεν όσον αφορά το επόμενο κολέγιο των ε, επιτρόπων. Ε, είναι γεγονός ε, ότι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελό μου είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι σημαντικά και όσον αφορά και τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Σκέφτομαι κυρίως τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια με τα οποία ήδη έχουμε κάνει τρομερές πρόοδους όσον αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο αλλά επίσης και τους εταίρους μας στην Αφρική. Έκτη πρόκληση αφορά τον πολιτισμό. Όπως κατεδείχθη στο Ευρωπαϊκό Έτος του 2018, ο πολιτισμός μας μέσα στην ποικιλομορφία του είναι αυτός ο οποίος μπορεί και πρέπει να καθορίσει τις κοινέ μας αξίες. Ε, κυρίως δε την ε, βούλησή μας να βάλουμε τον άνθρωπο ε, στο κέντρο όλης της, προσπάθειάς μας, της προσπάθειάς μας. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να υποστηρίξουμε την δημιουργικότητα των καλλιτεχνών μας και να προωθήσουμε την τεχνολογική καινοτομία ε, ακόμα και στον καλλιτεχνικό τομέα η έβδομη πρόκλησή μου είναι η δικιά σας, δηλαδή να διατηρήσουμε ε, την πρόταση όσον αφορά έναν ικανό προϋπολογισμό για όλους τους τομείς ε, την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Τέλος, η τελευταία πρόκληση που οπωσδήποτε δεν είναι η λιγότερο σημαντική είναι η θέση των γυναικών. Ξέρετε, ε, την άποψή μου για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι παραμένει και στη νέα μου θητεία ε, απαράλλακτη η θέση μου και η δέσμευσή μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω δεσμευτεί ενώπιόν σας να συνεχίσω ε, να βάζω τον πολίτη στο κέντρο της πολιτικής μου δράσης και ε, εδώ θα ήθελα μπροστά σας να, πάρω και μία, να αναλάβω και μία άλλη δέσμευση. Έχουν αλλάξει ε, οι καιροί. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Τα ατού ε, τα ισχυρά μας σημεία θα πρέπει να διατηρηθούν και τα ασθενή μας σημεία θα πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν ισχυρά. Θέλουμε να ξεφύγουμε από τις πεπατημένες. Θέλουμε να σκεφτούμε με τρόπο ε, διαφορετικό, ενδεχομένως ε, κάνοντας και ρήξεις. Θέλουμε να υφάνουμε ισχυρές, ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς τους αλαβάστρινους πύργους των θεσμικών οργάνων και θέλουμε να δημιουργήσουμε να συνδημιουργήσουμε όλοι μαζί, ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλοι οι πρωταγωνιστές το μέλλον μας. Με άλλα λόγια, δεσμεύομαι να φέρω την ε, καινοτομία ε, και την νεολαία στη δράση μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να στραφώ προς τους συναδέλφους Στου εκπροσωπού των πολιτικών ομάδων να πάρουν το λόγο και να σας υπενθυμίσω ότι έχετε ένα λεπτό για κάθε ερώτηση. Στη συνέχεια η κυρία Γκαμπριέλ θα έχει δύο λεπτά για τι απαντήσεις της. Αν θέλετε να κάνετε επερώτηση για το ίδιο θέμα, σας διατίθεται άλλο ένα λεπτό και άλλο ένα λεπτό θα έχει η κυρία Γκαμπριέλ για να απαντήσει. Η κυρία Σόντροβα, που είναι και συντονίστρια στην Επιτροπή Πολιτισμού και εκπροσωπεί το ΕΛΚ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Σόντροβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ συνοπτική απάντηση που δώσατε στι ρεπτέ μας ερωτήσεις. Σύμφωνο μαζί σας με αυτά που μας γράψατε. Ο πολιτισμός είναι στο DNA της Ευρώπης και η έρευνα και η εκπαίδευση πάνε χέρι-χέρι. Γι' αυτό το λόγο εμείς, ε, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και οι εμπειρογνώμονες αλλά και οι πολίτες αυτό που θέλουν να δουν στην πολιτισμό και την εκπαίδευση και την έρευνα. Ο τίτλος του χαρτοφυλακίου σας είναι καινοτομία και νεολαία. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για το μέλλον των πολιτών μας. Ο τίτλος, ωστόσο, δεν αποτυπώνει ωστόσο το, το ευρύ αυτό φάσμα του χαρτοφυλακίου σας. Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, νεολαία, αθλητισμός. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν ότι θα δώσετε σε όλους τους τομείς της πολιτικής την απαραίτητη, τη δέουσα προσοχή. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε τις βασικές σας προτεραιότητες ε, σε αυτό το τόσο ευρύ χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, η κυρία Γκάμπριελ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σοντροβά για τις ερωτήσεις σας. Όλες αυτές οι προτεραιότητες ε, ελπίζω να μπορέσω να σας παρουσιάσω στην Ακροασία. Όσο πιο πολύ σκέφτομαι στο περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου, κοιτώντα το θέμα τη καινοτομία και τη ανάπτυξη, την πολιτισμό, την νεολαία, επιτέλου όλα αυτά συνενώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο και βλέπω ότι είναι τεράστιε οι προκλήσει, αλλά υπάρχουν τεράστιε ευκαιρίε. Οι προκλήσει θα σα παρουσίασα. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ξεχωριστές εργασίες. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες και μιλώ σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμό. Θα πρέπει να υπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση προκειμένου αυτή να μας βοηθήσει και να φροντίσουμε στο επόμενο πλαίσιο η έρευνα να ενταχθεί σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Πώς όμως θα τα κάνουμε αυτό αν δεν κερδίσουμε την νεολαία, αν δεν έχουμε τις, αρμόδιες, τις κατάλληλες αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους νέους. Στο εξή λοιπόν θα ήθελα να ταχθώ σε αυτό το σκοπό. Θα ήθελα να εξετάσουμε τις ενδεχόμενες συνέργειες σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την νεολαία και την ε, αθλητισμό με την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό μας προσφέρει τόσες ευκαιρίες και μιλώ στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές συνεργίες στο Creative Europe σε ό,τι αφορά τις δημιουργικές βιομηχανίες και το δημιουργικό κλάδο. Επίσης, μεγάλη συνέργεια μεταξύ έρευνας, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα ήθελα να δώσουμε νέα πνοή σε αυτόν και στην καινοτομία σε ό,τι αφορά τον τρίτο πυλώνα θα ήθελα επίσης να με υπογραμμίσω τη νέα ιδέα να υπάρξει ένας χώρος εκπαίδευσης, ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης, γιατί θα πρέπει η διάσταση αυτή και η έρευνα να ενταχθεί στα πανεπιστημιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ορίσουμε λοιπόν τέτοιες προτεραιότητες στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Θα ήθελα αυτοί οι τρεις ε, τομείς που έχουν να κάνουν με διαφορετικές πτυχές ε, να τονιστούν ως υποδείγματα για τους πολίτες στα πλαίσια του εκπαίδευσης και του πολιτισμού να δώσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν τους νέους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να προσθέσω ένα θέμα, ένα ερώτημα για τον προπολογισμό. Ξέρετε το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το Erasmus και το Erasmus Plus για τη νέα περίοδο. Πώς θα γίνει αποτελεσματικό το πρόβλημα με νέες πρωτοβουλίες για να υποστηριχθούν από αυτά τα κονδύλια. Διότι είναι κρίσιμα προγράμματα για τους φοιτητέ, για τους σπουδαστέ σε επαγγελματική κατάρτιση και για τους καθηγητές. Πώς λοιπόν θα προκύψει ή θα καταφέρετε να πετύχετε αυτή την αύξηση των αναγκαίων πόρων. Η κυρία Γκάμπριλ απαντά. Εγώ υποστηρίζω το τυπεσιασμό ε, του προπολογισμού όπω το ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο και όπω δεσμεύτηκε να το εφαρμόσει η εκλεγήσα σαν πρόεδρος του, του, της Αφού θα πρέπει να συναντήσω με του υπουργού παιδεία για να... Και πριν συζητήσω με του υπουργού παιδεία, πρέπει να συζητήσω με τους υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, και για την έρευνα και την εντομία και για τον ορίζοντα Ευρώπη και για το πρόγραμμα Έρασμος πρέπει να πείσουμε εκείνου που θα λάβουν τις αποφάσεις την τελική απόφαση για να μας υποστηρίξουν. Όσον αφορά το πρόγραμμα Έρασμος, είναι ένα σύμβολο, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τώρα θα πρέπει να καλύψει ευρύτερο τομέα. Θα δρομολογήσει όλα τα μέτρα που θα καλύπτουν περισσότερους. Και για την, για την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, για τους καθηγητές. Όσον του καθηγητές, εγώ θα επέμενα επί τους καθηγητές γλωσσών. Διότι σήμερα χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Μια κινητικότητα της δύο του έρασμος αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Θα πρότεινα και ένα πράσινο έρασμος. Η νεολαία μας μας έστειλε, πιστεύω, ισχυρότατο μήνυμα. Το περιβάλλον, αλλαγή συνηθιών απαιτείται, χρειάζονται δράσεις και αυτή είναι μια συγκεκριμένη ιδέα που εκφράζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νίκα ο οποίο είναι συντονιστή από Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε για την Επιτροπή Βιομηχανία Ήτρε. Έχετε λοιπόν ένα λεπτό, κύριε Νικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία υποψήφια επιτροπέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Μία ερώτηση να σα κάνω συγκεκριμένη. Αν υπάρχουν διαφωνίε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τον προπολογισμό για τον Horizon Europe, ποιο θα υποστηρίξετε, το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ο οποίος, το οποίο Συμβούλιο μάλλον θα προτείνει λιγότερα χρήματα. Και το θέμα του μη συγχρονισμού των προτάσεων για τον προπολογισμό, πώς θα το λύσετε. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ε, επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί. Κάτι ακόμα. Μία ερώτηση ακόμα να σας κάνω. Τα έργα για την αξιολόγηση, πώς θα τα ε, ε, υλοποιήσετε το 2020 ή αργότερα για την έρευνα. Και εδώ έχω ένα πρόβλημα να επισημάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει σε εμπορική αξία τα προγράμματα έρευνα. Αυτό πώ θα το επιλύσετε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία και για του πολίτε αλλά και για την οικονομία. Γιατί έχουμε εξαιρετική έρευνα προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τον ε, προϋπολογισμό, εγώ ε, συμπορεύομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποστηρίζω ε, με ρόμοι την αύξηση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για το Horizon είναι επένδυση και όχι δαπάνη. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, ε, την ε, ψηφιακή ε, τροποποίηση και γενικώ τέτοιου είδους συνολικές προκλήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. 33% των θέσεων εργασίας έχουν δημιουργηθεί ακριβώς λόγω της εντατικοποίησης της γνώσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και αναφέρομαι στη φωνή του Κοινοβουλίου και επιτρέψτε μου να πω ότι ε, η κοινότητα των επιστημόνων, των ερευνών θα πρέπει να έρθουν μαζί μας έτσι ώστε η φωνή μας να γίνει πιο ε, δυνατή. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι παραμένοντας ρεαλιστές. Ε, όσον αφορά ε, τις αποστολές και τις εταιρικές σχέσεις, όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο πάντα ήταν μέρος της συζήτησης. Κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμφωνήσουμε μαζί σας ότι ας πούμε η νέα αρχή για τις εταιρικέ σχέσεις, η νέα προσέγγιση είναι να επιβάλλουμε επιμείνουμε ε, στο άνοιγμα, τη διαφάνεια και την προστιθέμενη αξία, θα έχουμε την δυνατότητα να μιλούμε με μία ε, φωνή. Θέλω λοιπόν να συνεργαστώ στενότατα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα περιμένω ας πούμε να αρχίσουν οι αποστολές το 2021 έτσι ώστε να ενημερώσω το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν πρότεινα ε, στα Mission Boards το κάθε Mission Board να ορίσει και ένα μέλος του Κοινοβούλιο έτσι ώστε ε, να μπορεί να ενημερώνει κάθε φορά ποιες είναι οι αποφάσεις και ποιες είναι οι εξέλιξεις. Πρώτο ε, πιλωτικό είναι το 2020, αλλά πραγματικά θα ήθελα πρώτα ε, να μιλήσω με την ομάδα μου. Δεν θέλω να τους δημιουργήσω πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκα για επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ. Είπατε ότι θα συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Ε, δεν, μας, ε, ε, θέλουμε να μας πιάνετε εξαπίνης, θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Η δεύτερη ερώτηση λοιπόν, πώς θα οργανώσετε τον διάλογο με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε από κοινού τα καλύτερα αποτελέσματα και έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε από κοινού τις ευέλτιστες ε, ε, αποφάσεις. Και περιμένω ακόμα ερώτηση, απάντηση συγγνώμη για την τελευταία μου ερώτηση. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει έρευνα προχωρημένη στην Ευρώπη αλλά ο καρπός της έρευνας δεν βρίσκεται στην αγορά της Ευρώπης. Απάντηση. Όσον αφορά το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά πιστεύω ότι ήμουν πολύ σαφής. Θα είναι ένας ε, ε, ισχυρός διάλογος και θα ξεκινήσει ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει να στραφεί κανείς στα όσα έχουμε προβλέψει στο Horizon Europe και στο 2020. Αν θέλουμε να περάσουμε αυτό το βήμα, όταν θέλουμε δηλαδή το αποτέλεσμα τη έρευνα με τα μετασχηματιστεί σε προϊόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις αποφάσεις. Αυτό γίνεται πλέον με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, καινοτομία. Θα πρέπει να συνεχιστεί. Ε, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε, ε, όπως είπα και προηγουμένως, οι ε, ε, μελετητές μας, οι ερευνητές μας να είναι καινοτόμοι και η καινοτομία να βασίζεται στην έρευνα. Σκέφτομαι ας πούμε στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αποστολές ναι, γιατί βεβαίως ε, θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι όλα αυτά ε, που γίνονται για αυτούς είναι απαραίτητα και ωφέλιμα. Ε, τώρα, για να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα, θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη εκστρατείας πληροφόρησης. Ε, η επιστήμη θα πρέπει να συναντήσει τους νέους, η επιστήμη θα πρέπει να συναντήσει ε, τους ε, πολίτες. Γι' αυτό υπάρχουν οι πρωτοβουλίες Science Meet Regions, Science Meet Young People κτλ. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήσαμε περισσότερο χρόνο γιατί ήταν πιο σύντομος ο κ. Νίκα η κυρία Φάρακ, συντονίστρια της, από την ομάδα Renew της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργισμού. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού μας χώρου χρειάζεται καινοτομία και χρειάζεται και συνέστημα. Ο πολιτισμός, τα μνημεία μας, η ιστορία μας συμμετέχουν σε αυτό. Να θυμηθούμε και την πυρκαγιά της Νότρο Ντάμ των Παρισίων που το έδειξε αυτό. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση για την ευρωπαϊκή αυτή κληρονομιά που επηρεάστηκε πολλές αλλαγές και από αυτούς που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Η ευρωπαϊκή κληρονομιά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ευρωπαϊκές πολιτικές. Και πρέπει να είναι πολύ σχεδής η προσέγγιση. Πρέπει να εμπνέεται από το παρελθόν και να προβάλλει στο μέλλον. Η προστασία της κληρονομιάς, η ορατότητα, η προσβασιμότητα, η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσία, γνώσης και κινητικότητα των ειδικών και για των καλλιτεχνών για να σχετίζεται ε, η κληρονομιά του παρελθόντος με τη νέα τεχνολογία και την κίνηση προς το μέλλον. Πώς μπορείτε όλα αυτά να τα διαθρώσετε, να συγκεράσετε αυτές τις προκλήσεις και τις ε, δυνατότητες που προσφέρονται, τόσο ώστε να προβάλλετε και στο μέλλον αυτή την κληρονομιά και να την προστατεύσετε. Για την ερώτησή σας, συμμερίζομαι απόλυτα αυτή την άποψη. Η πολιτισμική κληρονομιά είναι κάτι που είναι μοναδικό. Αν δούμε την επιτυχία που είχε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς με δεκάδες χιλιάδες ε, εκδηλώσει, με συμμετοχή εκατομμυρίων ατόμων. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να θέσουμε το ερώτημα πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό, ε, να εξασφαλίσουμε μια εξέλιξη σε σχέση με τα γνωστά. Γι' αυτό τη στιγμή του Ευρωπαϊκού Έτους τη πολιτιστική Κληρονομιάς είχαμε απίστευτο δίκτυο που δημιουργήθηκε από το τοπικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ, ένα βήμα για την πολιτιστική κληρονομιά, για την κληρονομιά μα αυτή. Θα συνεδριάσει για πρώτη φορά 15 Οκτωβρίου και θα καλούσε εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσέλθει, να συμμετάσχει στι συζητήσει για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη βάση συζητήσεων που θα δημιουργηθεί και τι δρόμου θα δούμε. Και θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί επίση η πολιτιστική μα κληρονομιά. Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Τη στιγμή της τις ημερίδες το Digital Date 3, ε, συζητήσαμε την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λιγότερο από 10% έχει ψηφιοποιηθεί σήμερα και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες μαζί με τα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, προφανώς θα ήθελα να αναφέρω ε, ότι είχαμε πολλές καλές πρωτοβουλίες μαζί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει αυτός ο χώρος να γίνει πιο ελκυστικός για τους νέους, πιο ελκυστικό για εκείνου που δεν έχουν πρόσβαση, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στον πολιτισμό σε περισσότερου ανθρώπου, Διότι όταν δούμε τι γίνεται, το 1 τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών λέει ότι δεν συμμετέχει σε πολιτιστικέ δραστηριότητε. Αυτό με τρομάζει σαν αριθμό. Θα επιμένω από τούδε και στο εξή, στι δράσει για την πολιτιστική κληρονομιά στον πρώτο πυλώνα, να ενισχύσουμε τη συμπερίληψη περισσότερων μέσω ψηφιοποίηση και μέσω νέων συνεργασιών τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό κεφα... Ε, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα καινοτομίας. Όταν βλέπουμε τις υποψηφιότητε, οι περισσότεροι ε, πρότειναν προγράμματα που δίνουν προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ και ξέρω ότι είναι στενά τα χρονικά όρια και έχετε πολλά να πείτε. Ε, περώτηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Να επανέλθω στο θέμα της ψηφιοποίησης, την οποία και αναφέρατε. Αυτό που με ανησυχεί σε ό,τι αφορά τη χάραξη του χαρτοφυλακίου είναι ότι ο πολιτισμός και η ψηφιοποίηση και η ψηφιοποίηση όπως είπατε έχει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα του πολιτισμού και έχω υπόψη μου και τις ευκαιρίες που έχει να προσφέρει σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης ε, Δυστυχώ αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην επιστολή αποστολή σα. Ο ρόλο σα ποιο θα είναι, ποια θα είναι η σχέση σα ε, τη κυρία Ελβί Γκουλάρ, που είναι υποψήφια επίτροπο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό της, ε, του πολιτισμού, πέρα από τα δίκτυα, πέρα από τη βιομηχανική, αν θέλετε, πτυχή αυτή, την πτυχή ανάπτυξη. Δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει μια πολιτική όπω όλε οι άλλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκάμπριελ, για να απαντήσει. Αυτό γίνεται ήδη στο τρέχον πρόγραμμα Creative Euro. Ήμουν υπεύθυνη για προγράμματα μέσα και ο να Ναύρατσης ήταν υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού. Αυτό δεν εμπόδισε την καλή συνεργασία. Αυτό λοιπόν βάσει τη εμπειρία μου ε, μπορώ να σα πω ότι η εμπειρία μου μου έδειξε ότι μπορούν να υπάρξει στενή συνεργασία και με την κυρία Γκουλάρ συνέργειες. Λοιπόν, μέσα στο χαρτοφυλάκιό μου υπάρχουν πολλές τέτοιες συνεργασίες σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Να μην ξεχνάμε ότι στο επόμενο Horizon Europe, στο δεύτερο πυλώνα, έχουμε μεγάλες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα του πολιτισμού, αμα, της ε, συμπεριπτικής κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να δοθούν σε αυτό το πλαίσιο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια της καινοτομίας τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Creative Europe. Πώς θα υπάρξουν συνεργασίες. Όλα αυτά αγγίζουν τον τομέα των μέσων ενημέρωσης και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε χάρη στην ανάπτυξη την ψηφιακή, νέες μορφές επικοινωνίας αναπτύχθηκαν. Αυτό προφανώς δεν είναι μόνο ευκαιρίες, έχει και απειλές τίθεται το θέμα α, το copyright. Ξέρουν οι δημιουργοί σε τι αναφέρομαι. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να οριστούν, να οριστούν οι προσανατολισμοί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακοπτή ο Πρόεδρος και νομίζω ότι υπάρχουν α, και άλλα θέματα τα οποία δεν απαντήσατε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο στο τέλος των παρεμβάσεων σας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητή είναι η κυρία Γενμπού, η οποία είναι συντονίστρια από την ομάδα των Πρασίνων στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρία Γκαμπριέλε. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε μία Ευρώπη, ούτε έναν τρόπο ζωής, ούτε μία κουλτούρα. Στην ε, γραπτή σας απάντηση μας είπατε ότι ε, η Ευρώπη θέλει να αναδείξει ε, αυτήν αυτόν τον πλούτο. Ξέρουμε πάντως ότι υπάρχουν κάποιες, κάποιοι πολιτισμοί οι οποίοι είτε προέρχονται κυρίως από τη μετανάστευση είτε από παλιά πολλές ε, απικίες ε, που πραγματικά ε, υποβιβάζονται. Επίσης πολιτισμοί των υπερποντίων διαμερισμάτων κλπ. Πώς θα κινηθείτε έτσι ώστε όλοι αυτοί οι πολιτισμοί, όλες αυτές οι κουλτούρες να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επίσης θα έχετε κάποιο πρόγραμμα έτσι ώστε τα λησμονημένα εδάφη να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η πολιτιστική πολυμορφία είναι ε, πραγματικά ε, η πηξίδα που μας οδηγεί σε οποιασδήποτε αποφάσεις παίρνουμε. Ε, το ίδιο συμβαίνει και τώρα στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους. Εκεί υπάρχουν προγράμματα τα οποία δουλεύουν ακριβώς για τις μικρές γλώσσες, τις περιφερειακές γλώσσες, τους μικρούς πολιτισμούς ε, ε, ε, πραγματικά έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη βοήθεια από τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κανείς να βρει στοιχεία απάντησης και να δεχτούμε όλοι ότι μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να αγγίξουμε περισσότερους πληθυσμούς. Επίσης, η διεύρυνση του προγράμματος Έρασμους είναι πάρα πολύ σημαντική αποφασίσαμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα και με πιο μικρές ε, οργανώσεις ε, έτσι ώστε μικρότερες οργανώσεις να έχουν την ε, δυνατότητα να επιλεγούν. Επίσης, μέσω του κεφαλαίου του αθλητισμού μπορούμε ε, να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, γιατί έχουμε δει ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι αποτελεσματικός και όσον αφορά την ενσωμάτωση μεταναστών και όσον αφορά την συμπερίληψη νέων που κινδυνεύουν να ριζοσπαστικοποιηθούν ή να απομακρυνθούν από τις δομές. Στο νέο πρόγραμμα Έρασμους λοιπόν θα πρέπει να εντάξουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και τέτοιου είδους δράσεις. Ε, και μάλιστα εγώ θα αναφερθώ σε μια ισομερή πρόσβαση για όλους. Ε, θέλουμε ε, να στείλουμε συγκεκριμένα μηνύματα. Στείλαμε άλλωστε συγκεκριμένα μηνύματα. Τώρα θα πρέπει να αποκτήσουν περιεχόμενο τα μηνύματα αυτά. Δεύτερη ερώτηση, συμπληρωματική. Κατάλαβα ότι συμφωνείτε με τον ευρωπαϊκό πολυπολιτισμό. Ε, πώς θα το συντονίσετε με την, ε, το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Σχοινά ε, που υπονοεί ότι υπάρχει ένας και μόνο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής του οποίου θα πρέπει να υπεραμεινθούμε και θα πρέπει να το προστατέψουμε. Απάντηση κυρία Γκαμπριέλ. Σε γενικές γραμμές εγώ δεν ε, ε, θέλω να αναφέρομαι σε διάφορους σεισμούς όπως ε, κουλτουρισμούς και τέτοιου είδους αφορισμούς. Nous avons ici des πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις συμπεριληπτικές ε, που θα έχουν στόχο όχι τόσο να προστατέψουν με αρνητική έννοια ή αρνητικό συνειρμό ε, κάποιες κοινότητες, αλλά να επιτρέψουν στις κοινότητες αυτές να αισθανθούν ότι συμμετέχουν ισότιμα. Αυτού του είδους τη συμμετοχή προσδο... Ε, περιμένουν και σε αυτή την συμμετοχή προσδοκούν οι νέοι μας. Υπάρχουν προγράμματα. Αναφέρομαι ας πούμε ε, στο Ευρωπαϊκό ε, Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, αναφέρομαι σε αυτούς τους νέους που ξεκινούν να βοηθήσουν μετανάστες, να βοηθήσουν παιδιά των Ρωμά και ταυτόχρονα να έχουν μια τρομερή εμπειρία Πρέπει να σας πω ότι πάνω από το 70% των συμμετεχόντων στο Erasmus λένε ότι μέσω του προγράμματος συνειδητοποίησαν ε, ότι δεν υπάρχει ένας πολιτισμός ή μία κουλτούρα ε, και νομίζω ότι μέσα από την κατανόηση θα αρθούν και οι παρανοήσεις. Ο κύριος Μπούκερ έχει το λόγο για ένα λεπτό από την Ήτρα. Κύριος Μπόρκα. Είμαστε σε παγκόσμια κλίμακα πρώτοι στην παραγωγή. Περίπου 162 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω και πάνω από μισό εκατομμύριο θέσει εργασία ε, δημιουργούνται από τον δημιουργικό τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει μεγάλο μερίδιο τη παγκόσμια αγορά για τα ελικόπτερα που πολλούνται στον κόσμο. Αν θα προστατεύσουμε τι ευρωπαϊκέ θέσει εργασία πρέπει να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες τεχνολογικές προκλήσεις, κυρίως για τη μείωση εκπομπών. Για να διαφυλάξουμε την ανωτερότητά μας την τεχνολογική, χρειάζονται οικονομικοί πόροι, επαρκής, για έρευνα όσον αφορά το μέλλον της, των αερομεταφορών με καθαρή, με λιγότερες εκπομπές. Θα δεσμευτείτε να εξασφαλίσετε ότι ο τομέας θα έχει την αναγκαία οικονομική υποστήριξη για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κόσμο, το τομέα της αεροναυτιλίας. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικός τομέας λοιπόν οι αεροπορικές μεταφορές και χάρη στην καινοτομία και την έρευνα μπορούμε να κάνουμε πρόοδο για να γίνει ο τομέας ε, πιο πράσινος. Και εδώ αναφέρομαι ήδη στην ιστορία που έχει το πρόγραμμα Clean Sky είναι ένα πρόγραμμα που μας επέτρεψε να κάνουμε πραγματική πρόοδο. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι στη δεύτερη φάση του τώρα και έχει σαν στόχο, χάρη στην καινοτομία, με τα νέα αεροσκάφη να μειώσουμε κατά 20 με 30% τις εκπομπές. Λοιπόν, θα ήθελα να τα θέσουμε όλα αυτά σε ένα πλαίσιο. Οι αερομεταφορές στα πλαίσια του Clean Sky 2 Λοιπόν, είναι θεσμική συνεργασία. Άρθρο 185 και 187 των συνθήκων οδηγεί σε αυτή τη συνεργασία και κάνουμε αξιολόγηση των συνεπιών των προγραμμάτων. Θέλουμε μέχρι το τέλο του έτου να έχουμε αποτελέσμα την έρευνα που διεξάγεται. Και σας διαβεβαιώ, καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς το Κοινοβούλιο να μπορεί να επιληφθεί και να ενημερωθεί. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να θυμηθούμε ότι οι συνεργασίες που θέλουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα, να έχουν αποτελέσματα οι συνεργασίες. Να είναι συνεργασίες που είναι σημαντικές για όλους και θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις. Δεν μπορώ να προδικάσω τελική απόφαση, αλλά πράγματι πρέπει να επιβεβαιώσω ότι οι αερομεταφορές εντάσσεται στη συνεργασία που προτείνεται και να συνεχιστεί αυτό και στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπόρκια. Διευκρινιστική ερώτηση. πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που θα καταβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προώθηση της υψηλής τεχνολογίας και στο ρόλο που θα παίξει αυτή η τεχνολογία. Απάντηση. Δίνω ιδιαίτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην καινοτομία, στο επόμενο πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Ήδη στα πλαίσια του παρόντος, του ορίζοντα 2020, έχουμε ένα καθεστώς χρηματοδοτήσεως κυρίως των μικρομεσών επιχειρήσεων. Έχουμε και άλλα μέσα και εργαλεία για την υποστήριξη αυτών. Θα τις βοηθήσουμε για να συμμετάσχουν σε διάφορες συμπράξεις και μέσω του ορίζοντα επιχειρήσεις Ευρώπης να ετοιμάσουμε διάφορε προτάσει. Στο επόμενο πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα είναι προνομίουχο στόχο στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα που είναι η Ευρωπαϊκή Καινοτομία. Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομία, αυτή είναι η φιλοδοξία μα. Δημιουργηθεί ενία θηρίδα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Για να μπορέσουν έτσι να μα προτείνουν προϊόντα, ιδέε, ρηξικέλευτε και να συνοδεύονται αυτέ και να διατίθενται στην αγορά πιο γρήγορα, να υλοποιούνται. Θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε άλλε δραστηριότητε, όπω το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία, έχω υπόψη μου τώρα, και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων φορέων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζενόφσκι, ο οποίο είναι συντονιστή από την ομάδα ECR στην Επιτροπή Γητρέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα ξεκινήσω, κυρία Γκάμπριελ, δίνοντα σα συγχαρητήρια για την υποψηφιότητά σα και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σαφή εκτίμηση της σκληρής δουλειάς και της εξαιρετικής δουλειάς που κάνετε στην προηγούμενη θετία. Η ερώτησή μου, στη διαπραγμάτευση του ορίζοντα Ευρώπη, εγώ και οι συνάδελφοί μου καταφέραμε να βάλουμε την αναφορά σε αυτό που ονομάζουμε τη μεταμόρφωση των περιφερειών, το οποίο θα υπάρξει σε ό,τι αφορά την υψηλή κατανάλωση του άνθρακα. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι η επιστήμη και η έρευνα έχει να σχετιστεί με τη μεταμόρφωση αυτή, με τη μετάβαση αυτή την οποία χρειάζεται η Ευρώπη. Θα υποστηρίξετε τέτοιου είδου προγράμματα σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σα σχέδια και τα σχέδια δράση σα. Η απάντηση είναι ναι, θα υποστηρίξω τέτοια έργα και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Στις περιφέρειες ε, όπου υπάρχει αυτή η μετάβαση. Είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτή την πρόκληση ήταν να αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Να μειώσουμε τη διοξίδη του άνθρακα, τι εκπομπέ του διοξίδη του άνθρακα σε ό,τι αφορά και τον ορίζοντα 2020. Επενδύσαμε σε τεχνολογίες για την αποθήκευση, την α, χρήση του διοξιδίου του άνθρακα προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Η τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει ε, να προχωρήσει γιατί χωρίς ε, την έρευνα και την ανάπτυξη δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις περιφέρειες. Γιατί εδώ θα θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Έχουμε σαφείς πολιτικές φιλοδοξίες σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Έχουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε για να τους πετύχουμε. Μία πολιτική φιλοδοξία δεν μπορεί να είναι εις βάρος της ε, κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχω υπόψη μου όλους όσους ζουν σε τέτοιες περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν είναι τεράστιε αυτέ οι προκλήσει και σχετίζονται με άλλα τμήματα του χαρτοφυλακίου. Πώ θα φροντίσουμε να έχουν εργασία και να έχουν απαραίτητε ικανότητε και δεξιότητε αυτοί οι άνθρωποι, να είναι ανταγωνιστικοί. Ναι, θα υποστηρίξω τι πρωτοβουλίε αυτέ. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο λεπτομερώ. Ah, είχατε χρόνο, είχατε χρόνο, λέει η Πρόεδρο. Συγγνώμη, είχαμε βάλει το ο χρόνος στο ένα λεπτό. Να συνεχίσω λοιπόν, λέει η κυρία Γκαμπρίλ, για να ολοκληρώσω. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν, γιατί αναφέρεστε στην μετάβαση. Να σας υπενθυμίσω όμως καταρχάς ότι έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η μετάβαση όχι μόνο στην έρευνα και στην οριζοντά 2020 αλλά και με την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από τον ε, Αντιπρόεδρος Εύκοβιτς, ε, για να ε, συνενωθούν αυτές οι περιοχές οι οποίες πλήττονται και προκειμένου να ληφθούν κοινέ αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μου. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές, να δώσουμε αρμοδιότητες. Εδώ η κατάρτιση και η εκπαίδευση θα έχουν βασικό ρόλο. Η εκμάθηση λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι περιφέρειες να υπολογίζουν του πόρου που έχουν για να μην χάσουν την ανταγωνιστικότητά του. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο, ο κ. Σανόφσκι να κάνει την επόμενη ερώτηση, αν θέλει. Ναι, μια διευκρινιστική ερώτηση για τον ορίζοντα Ευρώπη, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία. Σε τι βαθμό σκοπεύετε να υποστηρίξετε το προγράμματα για το διάστημα Γαλιλαίο, NGONOS, Κοπέρνικος, που αποτελούν, αν θέλετε, μια φανταστική ευρωπαϊκή ιδέα, μια τεράστια ευκαιρία για τις νεοφύσεις εταιρείε για τους ε, νέους. Μια εξαιρετική λοιπόν ευκαιρία για το μέλλον. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη μπορεί να είναι περήφανη, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρώπης. Το διάστημα και οι υπηρεσίες διαστήματος είναι πολύ κεντρική σημασία για την Ευρώπη. 10% του ΑΕΠ τη Ευρώπη έχει να κάνει με τις διαστημικέ αυτές υπηρεσίε. Είπατε, το, αναφέρατε τον Κοπέρνικο, το Γαλιλαίο. Μεγάλε ιστορίε επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καταδεικνύουν ότι είμαστε δυνατοί. Είμαστε σε θέση με τι επένδυσεις που έχουν γίνει στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και στον οριζοντά να πετύχουμε πραγματικέ επιτυχίε. Θα ε, υποστηρίξω λοιπόν τα προγράμματα αυτά. Είναι τεράστιο το δυναμικό επιτυχία τους και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, αλλά κυρίως επειδή οι υπηρεσίε αυτές για το διάστημα μας ανοίγουν ε, νέες, ε, νέα πρόσβαση σε ό,τι αφορά διάφορες εφαρμογές. Για παράδειγμα, η γεωργία με μεγάλη ακρίβεια. Εδώ μπορεί να μας βοηθήσουν οι υπηρεσίες για το διάστημα. Και επίσης σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των καταστροφών και εδώ είναι πολύ σημαντικό το σκέλος αυτός. Και ξέρετε ότι είναι στο χαρτοφυλλογείο της κυρίας Γκουλάρ, αλλά από την άλλη θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά σε διαφορετική προκειμένου αυτή η πολιτική να δημορφωθεί με πιο μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματίας, συντονίστρια της ΓΚΟΕ στην Επιτροπή Ήτρε. Κυρία Ματίας, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία υποψήφια επίτροπε. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις να σας θέσω. Καταρχάς, στον ορίζοντα Ευρώπη αναφέρατε ήδη ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε συμμετάσχει πλήρως πάντα στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε τα θέματα τεχνολογίας και στρατηγική καινοτομία. Η πρόταση όμως δεν έχει δώσει τα κατάλληλα μέσα να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άμεσο ερώτημα λοιπόν. Όσον αφορά αυτό, θα αποσύρετε αυτή την πρόταση και θα υποβάλλετε νέα πρόταση, η οποία θα δίνει στο Κοινοβούλιο ε, τις σωστές εξουσίες που θα πρέπει να διαθέτει ως συνομοθέτης. Δεύτερον, η προστασία των επιστημόνων και η πρόθεση και η ενίσχυση των επιστημόνων. Δηλαδή στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα. Τι εγγυήσει θα δοθούν για αυτό το τομέα. Να μην υπάρχει ένα μπλοκάρισμα κάποια σημαντική έρευνα, Φερρυπίν. χωρίς να έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιηθεί και να προωθηθεί. Ευχαριστώ. για τις ερωτήσεις κυρία Ματίας. Έδωσα κάποιες απαντήσεις, αλλά θα ήθελα το Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως στα βασικά σημεία, στο στρατηγικό σχέδιο και τις συνεργασίες και τη διεθνή συνεργασία. Είναι σημαντικότατο για μένα, όπως είπα, να σας ενημερώνω. Υπενθυμίζω ότι όταν θα μιλήσουμε για το στρατηγικό αυτό σχέδιο, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει μαζί να εντοπίσουμε αυτά τα προγράμματα που θα δώσουν τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την ευρωπαϊκή, τα προγράμματα που θα ανταποκριθούν στι προκλήσει, όπω είναι το κλίμα ή ο ψηφιακό τομέα, η ψηφιακή εποχή. Σα διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνω απολύτω στη διάθεσή σα. Αλλά θα, στις διαβουλεύσεις θα φροντίσω να λάβω υπόψη αυτά που είπατε όσον αφορά την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Ξέρετε γιατί προτείναμε το Euricast. Θέλαμε σαφήνεια και ορατότητα. Το Ινστιτούτο ανήκει στον ορίζοντα 2020 και στον ορίζοντα Ευρώπη θα ανήκει στο μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμαστεί. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τελευταία στιγμή. Ήδη τροποποιήθηκε σημαντικά ο τομέας το 2013 και νέε αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν. Να Εξασφαλίζεται η μετάβαση ευέλικτη προ τα νέα προγράμματα, Προ το νέο πρόγραμμα. Δεν θέλω να προδικάσω την απόφαση, ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια του προγραμματισμού για το νέο σώμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια χαρτοφυλάκια μπορούν να παραμείνουν όσοι έχουν προταθεί να αποσυρθούν και πρέπει να σεβαστούμε πλήρω το ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο ρόλο των συνομοθετών. Ουσιαστικά, αυτό είναι που σημαντικό για μένα, είναι να παραμείνω στη διάθεσή σα και σα διαβεβαιώνω ότι θα συνεργαστώ μαζί σα στενά για να βρούμε έναν ε, κανονισμό που θα επιτρέπει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συντούτο Τεχνολογίας να ε, συμπληρώσει το τρίγωνο της έρευνα καινοτομία ε, και της καινοτομία. Λοιπόν, όσον αφορά τι πτυχέ τι κοινωνικέ, θέλουμε όλε οι πτυχέ των ορίζοντα Ευρώπη να λαμβάνονται υπόψη και όχι μόνο ε, στι εκπομπέ, αλλά να μπουν και στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα. Θα ήθελα να μην απομονωθούν κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όταν θα προσπαθούμε να καινοτομούμε στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα ή όταν θα ε, πρέπει να κινηθούμε και να έχουμε προγράμματα στο δεύτερο πυλώνα. Επερώτηση για την κυρία Ματία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους ε, που έκαναν μια περώτηση που δεν είχε να κάνει απαραίτητα με το πρώτο σκέλος των ερωτήσεων και θα ήθελα να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σημείο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 136 αναφέρεται ότι καμία χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει στον τομέα της έρευνας αν ε, συνεπάγεται, ε, μάλλον αν είναι σε κράτος ε, που έχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου. Στον ορίζοντα 2020 μιλάμε για επενδύσεις σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, σε ό,τι αφορά στρατιωτικά στοιχεία. Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφύγουμε χρηματοδοσία, χρηματοδοσία χρήματα σε επιχειρήσεις που έχουν, ε, έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Η κυρία Γκαμπριέλα. ένας τρόπος μόνο υπάρχει η απάντηση. Να σεβόμαστε τα δεδομένα. Να βλέπουμε λοιπόν τις πληροφορίες ε, όταν κάτι δεν ε, πάει καλά. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το Μαρόκο που ρωτήσατε αλλά σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι αφορά την ε, αρχή της εδαφικότητας, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά επίσης ε, τη συνεργασία με τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες ε, του Ισραήλ που έχουν να κάνουν με θέματα πληροφορικής για τα είδατα και ούτω καθεξής. Γιατί πρέπει να φροντίσουμε όταν ε, δεν γίνουν σεβαστοί οι κανόνε σε έναν τομέα, να αποκλείεται η συνεργασία σε άλλου τομεί. Θα χρειαζόμουν πιο πολλέ ε, ε, λεπτομέρειε για τι υποθέσει που αναφέρετε και σας, να σα απαντήσω πιο λεπτομερώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Φερχάιεν για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Next speaker on our list is Mrs. Hanna Virkunen for EPP. Η κυρία Χένα είναι από το ΕΛΚ. Επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επιτροπέ. Ξέρουμε ότι το Horizon Europe είναι σημαντικό για την Ευρώπη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και την υλοποίηση ε, φιλόδοξων προγραμμάτων που δεσπίστηκαν ήδη στην προηγούμενη θητεία σας. Ε, ξεκινάει νέα συνεργασία ε, με και με όσους εφαρμόζουν ε, την διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ε, είπατε προηγουμένως ότι θα ζητήσετε τη συμμετοχή μας ε, σε ε, όσον αφορά τον σχεδιασμό, τις αποστολές κλπ. Οπωσδήποτε εμείς θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί μας όσο γίνεται περισσότερο. Είπατε ότι θα ξεκινήσετε κάποιες στενές σχέσεις και ίσως ε, τακτικές συναντήσεις με το Κοινοβούλιο, πάντα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Πώς έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε, ε, κυρία Γκάμπριελ. Στην ε, πράξη. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να ανταλλάσσουμε κάποια έγγραφα. Εγώ θα ήθελα να έχουμε τακτικές συζητήσεις με συγκεκριμένο θέμα και οι συζητήσεις μας να ακολουθούν ε, τα θέματα αυτά. Ας πούμε, μία φορά τον μήνα να ε, βλέπουμε πού έχουμε προχωρήσει και πόσο έχουμε προχωρήσει. Ε, η συμμετοχή θα μπορούσε να γίνει με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε, π.χ. συνάντηση με τους συντονιστές στο Στρασβούργο ή συνάντηση εδώ. Ε, επίσης θα ζητήσω και από τις ε, υπηρεσίες μου να ξεκινήσουν μια πραγματική εκστρατεία πληροφόρησης. Θα ήθελα να πάμε σε όλες τις χώρες να παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα εφαρμόζοντας όμως μια προσέγγιση αναχώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, ε, θα συζητώνται οι προκλήσεις και που αφορούν και την υλοποίηση των εταιρικών σχέσεων. Καμία απόφαση όμως δεν θα λαμβάνεται χωρίς πρώτερη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει λάβει γνώση. Αυτό τι είναι η θέση μου όσον αφορά τις αποστολές, όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις, ε, έτσι ώστε ε, πραγματικά ε, να λυθούν από κοινού ζητήματα τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε να προωθήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σωστότερα να, να προετοιμάσουμε την υλοποίηση. Έχετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση, ναι κυρία Πρόεδρε σχετικά με το Horizon Europe και τον προϋπολογισμό. Αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές ο προϋπολογισμός. Νομίζω πάντως ότι είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα για την Επιτροπή μας αλλά και για την Ευρώπη. Αυτό το θέμα δηλαδή της αύξησης του προϋπολογισμού του Horizon Europe ε, 120 δις ε, προϋπολογισμό έχει σκοπό το Κοινοβούλιο ε, να δώσει, αλλά βεβαίως τα ε, κράτη-μέλη είναι αυτά που παίζουν το σημαντικό ρόλο. Πώς εσείς προτίθεστε να πείσετε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν με αυτόν τον αυξημένο προϋπολογισμό. Είναι δύσκολη ερώτηση βέβαια και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 2015 ορίζον 2020 είχε περικοπεί 2 δις για την την θέσπιση του ε, Ταμείου στρατηγικών επενδύσεων και τώρα γίνεται μία προσπάθεια να πάλι να πάνε χρήματα και κονδύλια από αυτόν τον τομέα στο Invest EU. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ανεξάρτητος από τον προϋπολογισμό άλλων εργαλείων. Τι πιστεύετε εσείς κυρία Γκάμπριελ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος δεν θα επαναλάβω αυτά που έχω ήδη πει αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αν δεν κάνουμε τώρα επενδύσεις κινδυνεύει σε μερικά χρόνια η Ευρώπη να βρεθεί σε ένα σημείο χωρίς ε, επιστροφή. Ε, χάσαμε το προηγούμενο κύμα καινοτομίας αλλά θα πρέπει να αδράξουμε το νέο ε, κύμα καινοτομίας. Έχουμε απέναντί μας τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε ιστέρηση στέρηση ε, των ε, επενδύσεων στην ε, παιδεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν μιλάμε όμως για υστέρηση και στην έρευνα, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη επενδύει 217 εκατομμύρια στην έρευνα και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά πολύ κάτω από τον στόχο του 3%. Εγώ θέλω παραδείγματα ε, γιατί οι χώρες ε, οι οποίες έχουν ε, επενδύσει 3 έως 4% έχουν προχωρήσει πολύ και θέλουμε και σε άλλες περιπτώσεις να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας λόγω ακριβώς της έρευνας και της καινοτομίας. The next speaker... στον κατάλαβο είναι η κυρία mm. από Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στο μέλλον, ε, ε, στο μέλλον θα πρέπει να υποστηρίξετε τον ευρωπαϊκό κλάδο στον οποίο εντάσσονται και τα μέσα τα ακουστικά, τα οποία προφανώς και συνδέονται με τον πολιτισμό πολύ στενά. Τα προγράμματα του Creative Europe και ε, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ως τώρα έχει πάει πολύ καλά προς το παρόν. Έχετε δεσμευτεί και εσείς, αλλά αυτό θα είναι πλέον στο χαρτοφυλάκιο της Επιτρόπου για την Ιστορική Αγορά. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν ότι η Μελλοντική Επιτροπή θα συνεχίσει την πρόθεση των μέσων αυτών και θα τα θεωρήσει όχι μόνο από την οπτική γωνία της αγοράς, αλλά και από πλευράς του πολιτισμικού κλάδου, προκειμένου να υπάρχει σωστή υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ, η Επιτροπός Γκάμπριελ. σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, η συνεργασία ήταν ως τώρα άριστη. Το είπα και προηγουμένως αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει συγχρονισμός προφανώς των δράσεών μου με τους δράσεις της Επιτροπού Γκουλάρ. Σε ό,τι αφορά τον χρηματοδότηση του Creative Europe, δεν είναι τόσο μεγάλη η χρηματοδότηση. Από πλευράς μου όμως αυτό που θέλω είναι να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε ό,τι αφορά και τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Οριζόντας Ευρώπη. Έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια κοινωνία συμπεριληπτική στα πλαίσια του Οριζόντα Ευρώπη, σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, σε ό,τι αφορά την, τις απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα χάσματα που υπάρχουν, γιατί επαναλευθούν αυτές οι αδυναμίες το επαναλαμβάνουμε, δεν θα έχουμε την ευκαιρία αυτή. Θέλουμε να έχουμε κοινή δράση. Γι' αυτό λοιπόν για την κοινότητά της καινοτομίας και της γνώσης. Γι' αυτό λοιπόν το Σχετικό Ινστιτούτο έχει προβλέψει να υπάρξει μια νέα όθηση σε αυτές τις ε, πτυχές στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία στο μέλλον και με όσα έχουν ήδη γίνει στον ορίζοντα Ευρώπη. Αυτό θα αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει διαρκώς να είμαστε σε συνεργασία και σε συντονισμό μεταξύ μας για να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά που αναφέρατε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, το οπτικοακουστικά μέσα δεν θα παραμείνουν μόνο ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τα μέσα αλλά να συνταχθούν και να ενταχθούν σε ό,τι αφορά την έρευνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Κοινοτομίας και Έρευνας. Εγώ σίγουρα θα προσέξω ιδιαίτερα την, το σκέλος αυτός τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η έχετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση να κάνετε. Θα είχε νόημα ένα τέτοιο σχετικά μικρά, μικρό πρόγραμμα να μην το διαιρέσουμε περαιτέρω. Είπατε πριν από λίγο ότι θα είσαστε στην πλευρά, στο πλευρό του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης για τον ορίζοντα Ευρώπη. Ισχύει αυτό και για το Creative Europe, όπου το Κοινοβούλιο ζήτησε διπλασιασμό του πόρων και για το Erasmus Plus, όπου ζητήσαμε τριπλασιασμό της χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι απαραίτητο, γιατί ιδιαίτερα το Creative Europe είναι διαρκώς υποχρηματοδοτούμενο. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πολύ παραπάνω στόχους αν ε, είχαμε παραπάνω χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα που έχει πάρα πολλά καλά έργα να προσφέρει. Το ίδιο ισχύει και για τον ορίζοντα Ευρώπη. Είσαστε λοιπόν στο πλευρό του Κοινοβουλίου, θα προσπαθήσετε μαζί μας να πείσουμε το Συμβούλιο να διαθέσει πιο μεγάλη χρηματοδότηση προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι εν μέρη η απάντηση είναι σε αυτά που μπορούσα να κάνω τελευταία χρόνια. Θυμάμαι πολύ καλά στην, ε, όταν ήταν, μίλησα στην ακροσία μου για τα ψηφιακά, μίλησα ότι θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια των προγραμμάτων media, στα πλαίσια του Creative Europe. Είχα δει πολλά χαμόγελα τότε. Αυτό που πετύχαμε όμως ήταν 30%, 34% αύξηση ε, στην πρόταση που κάναμε. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να εξασφαλιστεί αυτό και μετά πραγματικά να φροντίσουμε μέσω συνεργασιών πόροι ίσως που δεν θα είχαμε σε αυτή τη φάση του Creative Europe να χρησιμοποιηθούν παρόλα αυτά, αλλά μέσω συνεργασιών με, εκείνα που, με εκείνους που προανέφερα. Έχουμε 52 δισεκατομμύρια στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα για τον ορίζοντα Ευρώπη, για τα clusters, για τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό, τη συμπεριληπτική κοινωνία. Θα υπάρξουν πολλά περισσότερα από τα 609 εκατομμύρια του τμήματος πολιτισμού του Creative Europe. Εγώ θα παραμείνω πιστή στην αύξηση που ζητήσαμε για να την εξασφαλίσουμε και μετά να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο μέσω άλλων προγραμμάτων όπως είναι αυτά που προβλέπονται στον ορίζοντα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ματίνα Γκλαμπάγιοβα, η οποία είναι συντονίστρια από το Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, χαίρομαι που το χαρτοφυλάκι όσα το βλέπετε σαν πρόκληση. Σίγουρα θα είναι. Είπατε ότι θέλετε να κάνετε τα πάντα για να υποστηρίξετε την τεχνογνωσία και το ταλέντο που έχουμε στην Ευρώπη και που έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για αυτά. Και αναφέρατε επίση ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι μεγάλοι φορεί που υποστηριχθούν, αλλά και οι μικρότεροι. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή οικονομία και παρόλο που θεωρητικά υποστηριζόταν, στην πράξη όμως πολύ συχνά μαθαίναμε ότι δεν γινόταν και πάρα πολλά. Όταν αναφερθήκατε στον τρίτο πυλώνα του ορίζοντα 2020, θα ήθελα να ξέρω τι άλλες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα βήματα θέλετε να λάβετε, προτίθεστε να λάβετε, πέρα από τα χρήματα που υποσχεθήκατε και πόσο προσωπικά, τι προσπάθειες θα καταβάλλετε για να ελοπίσετε τους στόχους σας. Καταρχάς, απάντηση. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν κάνουμε πολλά στον ορίζοντα 2020 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βέβαια και καλύτερα να τα πάμε. Αναφέρθηκα σε ένα αριθμητικό στοιχείο. Στον ορίζοντα 2020 στόχος για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν το 20%. Αυτό το ξεπεράσαμε κατά πολύ. Είμαστε πέρα από το 25%. Εγώ θα επέμενα και επί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη Καινοτομία. Ενία θηρίδα θα πρέπει να είναι όπου οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα έχουν πρόσβαση. Θα είναι βασική ομάδα στόχο. Έτσι δε περαιτέρω, διότι το Κοινοβούλιο υπήρξε σαφέστατο. 70% του προπολογισμού θα διατίθεται για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, για τι νέε επιχειρήσει. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να θέσω τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την υποστήριξη αυτών. Διότι ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομία. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ μπόρεσαν να διαθέσουν σε πάνω από 4.500 μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, γνωρίζουμε όλοι ότι θέλουμε αυτό να δημιουργεί επενδύσεις. Βλέποντας τα αριθμητικά στοιχεία στο 1 ευρώ που επενδύεται μέσω επιτάχυνσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παίρνουμε 2,34% απόδοση. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό που θα ήθελα να πω ε, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες θα πρέπει να είναι ενήμερες για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Θα πρέπει να έχουν πραγματική σαφήνεια μπροστά, να μην δημιουργούνται κλειστές λέσχες και γι' αυτό επίσης θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας, διότι και εκεί έχουν πρωτοβουλίες με στόχο την περιφερειακή καινοτομία. Επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σαν στόχο, αλλά ακούω όμως και τις κατηγορίες που ακούγονται για το πόσο κλειστό δεν υπάρχουν πολλέ δυνατότητες να έχουν πρόσβαση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όσον αφορά τις ε, ε, συγχρηματοδοτήσεις έχουν πρόβλημα. Θα θέλουμε όμως να καλύψουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά παντού στην Ευρώπη, να μην αφήσουμε καμία εκτός. Ευχαριστώ. Έχετε μήπως ευχαριστική ερώτηση. Ναι. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θα η υποστηρίξει τους καινοτόμους ε, ε, παράγοντες στην Ευρώπη, τις νεοφύης επιχειρήσεις για παράδειγμα. 70% λοιπόν του προπολογισμού θα πρέπει να ταχθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αν πιστεύετε, αν ε, λάβατε υπόψη ότι έχουμε 24 εκατομμύρια νεοφύης επιχειρήσεις, 28% δηλαδή, στο κλάδο, Άρκει το 70%. Και πώς ε, θα τις εισακούσουμε αυτές τις επιχειρήσεις ε, γιατί ξέρουμε ότι προτιμούν τις επιδοτήσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να τις εισακούσουμε και να γνωρίζουμε τι ζητούν και τι χρειάζονται. Η κυρία Κάπριελ. Νομίζω ότι ο προπολογισμό ποτέ δεν θα είναι αρκετό αν θέλουμε να απαντήσουμε σε όλε τι ανάγκε. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι σε συνέργειε και γι' αυτό αναφέρομαι και σε άλλε δυνατότητε που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ε, δεν θα υπάρχουν μόνο οι επιταχυντέ ή μόνο το Συμβούλιο ε, Καινοτομία, θα υπάρχει και το Invest EU. Θα υπάρξουν τεράστιε ευκαιρίε και δυνατότητε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να τα υποστηρίζουμε όχι μόνο για να ακούσουμε τις ιδέες όλων, αλλά και γιατί ε, θα μπορούμε να τροφοδοτηθούμε από αυτές ε, τις ε, ιδέες στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τις χρηματοδοτήσουμε έτσι ώστε να συμμετάσχουν, έτσι ώστε να ακούγεται η φωνή τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή σκέψεων, έτσι ώστε και ιδεών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ε, δικτύωση. Δεν υπάρχουν φυσικά ε, θαυματουργές λύσεις, αλλά από την άλλη μεριά να μην κλείνουμε την πόρτα σε άλλες δυνατότητες όπως είναι ε, το Invest EU και τις δυνατότητες που μπορούν να δώσουν και οι περιφερειακές συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Πίτερ Πόλακ, από την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και από το ΕΛΚΑ. Αξιότιμη κυρία υποψήφια Επιτροπέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά τα θέματα εκπαίδευσης. Μιλάμε για τρεις χώρες που διαχωρίζουν τα παιδιά Ρωμά σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν πρόκειται για παιδιά τα οποία σε σχολεία ε, συμμετείχαν μεν αλλά δεν είχαν ευκαιρίες ουσιαστικές σε μία χώρα. Ωστόσο πήγαν και στα πανεπιστήμια, έγιναν διευθυν... πήραν διευθυντικές θέσεις εδώ έχουμε ένα βασικό πρόβλημα λοιπόν, ένα θεμελιώδες πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τη γενικότερη ανάπτυξη της ε, χώρας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς σκοπεύετε τα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα να τα διαμορφώσετε με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δίρυβονται ευκαιρίε και στα παιδιά Ρώμα και να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασία στο μέλλον. Κυρία Γκαμπριέλ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σχετικά με τις ε, όσον αφορά συγκεκριμένα ε, τις όποιες διαδικασίες νομικές ε, έχουν ξεκινήσει σχετικά με διακριτική μεταχείριση, δεν θέλω να μπω ε, σε αυτές ε, τις λεπτομέρειες που αφορούν οπωσδήποτε ε, το χαρτοφυλάκιο της δικαιοσύνης. Βεβαίως θέλουμε τα παιδιά Ρωμά να συμμετέχουν στην πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται In School 31 σχολεία σε όλες τις χώρες που θα δημιουργηθούν έτσι ώστε όχι μόνο να γίνεται εστίαση καλύτερη στα παιδιά Ρωμά αλλά και αυτό είναι η καινοτομία ε, στα οποία θα δουλεύουμε περισσότερο με τις οικογένειες ε, και την κοινότητα ε, διότι η αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μόνο από την εργασία με τα παιδιά ή από το εκπαιδευτικό σύστημα προέρχεται και μέσα από την συνεργασία με την κοινότητα και με τις οικογένειες καθώς επίσης και με καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Εγώ θα παρακολουθήσω από κοντά αυτές ε, τις 31 ε, εκπαιδευτικές ενότητες για να δω ακριβώς πού μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί οπωσδήποτε αυτό θα αποτελέσει υλικό επί του οποίου θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω. Επομένως, ε, συμπερίληψη, πολύ σημαντικό στοιχείο, πολύ σημαντική λέξη, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεφύγουμε από τη λέξη και να έχουμε και περισσότερα προγράμματα, περισσότερες δράσεις τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Αξιότιμη κυρία Γκάμπριέλα. Η τα μέτρα για την κοινότητα των Ρωμά εφαρμόζονται εδώ και 20 χρόνια και εγώ προσωπικά έχω να πω ότι πολλά προγράμματα δεν είχαν οποιαδήποτε επιτυχία. Τα μέτρα λοιπόν αυτά, όπως σας είπα, ε, μιλάω για μία χώρα όπου τα παιδιά Ρωμά σημειώνουν επιτυχίες. Ενώ τα ίδια παιδιά δεν ε, μπορούν να πετύχουν κάτι. Το ερώτημα λοιπόν που σας απευθύνω είναι το εξής. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση σε κράτη-μέλη προκειμένου να μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα προκειμένου να μπορέσει κάθε παιδί να έχει ευκαιρίες επιτυχίας να μπορέσει να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαμπριέλα. Είπατε σωστά ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσει στα κράτη-μέλη και θα χρησιμοποιήσω τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα, λαμβάνοντα φυσικά υπόψη και τις αρμοδιότητές μας, σεβόμενοι τι αρμοδιότητε μα, Και μιλώ και για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πιστεύω ότι θα το πρέπει να το, χρησιμοποιήσουμε όλο και πιο πολύ και πιο συστηματικά στι συζητήσει με τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν συγκεκριμένε συστάσει με κατάλληλο τρόπο σε ό,τι αφορά τα εθνικά του συστήματα και λαμβάνοντα υπόψη τέτοιες, ε, τέτοια παραδείγματα αυτό λοιπόν που θα μπορούσα να κάνω είναι να αναφέρομαι συχνά στις συστάσεις ε, που διατυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να συνεχίζουμε να ευαισθητοποιούμε τα κράτη-μέλη, τηρώντας τις αρμοδιότητές μας. Αν δεν υπάρξει όμως ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα της συμπερίληψης, σε αυτό το θέμα που αφορά όχι μόνο τους νέους και τις επιχειρήσεις, πώς θα πετύχουμε πρόοδο στα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή είναι η Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ήτρε, η Πατρίτσια Τόγια από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Καλησπέρα κύριε υποψήφια επίτροπε. Είπαμε ότι θέλουμε ε, να βοηθήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις startups γιατί ξέρουμε ότι από αυτές πολλά προγράμματα έχουν εμπορευματοποιηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα μας διασφαλίσετε ότι δεν θα πέσουν σε αυτήν την αγχώνη, δεν θα περάσουν από αυτή την αγχώνη, από αυτή τη μου αυτά τα προγράμματα των καινοτόμων επιχειρήσεων. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει το δημόσιο χρήμα ε, να ε, λαμβάνει ε, η υπόψη όλες τις συνθήκες και να χρηματοδοτεί με όριμο τρόπο όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε τα προγράμματα να μην είναι απλά venture capitals. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και νέους και περισσότερους επιστήμονες και ερευνητές. Ποια θα είναι όμως τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιήσετε και επίσης τι είδους accountability ε, θα υπάρξει για τους αξιολογητές. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια. Ε, επιμένω λοιπόν και υπογραμμίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να, να εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα και την εμπορευματοποίηση. Ε, ε, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στη... στον επιστημονικό τομέα. πρόκειται μια πραγματικά πολύ σημαντική πρώτη ύλη, αλλά στην κοινοτομία υστερούμε. Γι' αυτό λοιπόν υπογραμμίζω ότι είναι απαραίτητη μια αλλαγή, μια τροποποίηση έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να δώσουμε, ε, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία ε, θα μπορούμε να τα βάλουμε στην αγορά. Ε, συνεργασία λοιπόν με τα πανεπιστήμια. Ε, έχουμε ήδη 17 ε, συμμαχίες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει με τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να προωθήσουμε την γνώση, να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε τα αποτελέσματα. Ε, με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό ε, και ξέρω ότι στις 12 Νοεμβρίου η Γενική Διεύθυνση Έρευνας ε, θα οργανώσει μία ημερίδα σχετικά, μία διάσκεψη σχετικά με την μετάδοση της γνώσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει μαζί με το Κοινοβούλιο να σκεφτούμε ποια είναι τα πιο επίγοντα μέτρα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την την ε, διαχείριση του προγράμματος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με τρομερές γνώσεις, κυρίως όσον αφορά την ε, τεχνολογία, τις νέες τεχνολογίες, αλλά οπωσδήποτε και αυτοί θα πρέπει να ε, είναι υπόλογοι και να αναφέρονται σε σχέση με την εργασία τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται και το Κοινοβούλιο για την πορεία της επιλογής των projects και της χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και να έχουμε ε, ε, εμπλουτισμό των επαφών και των γνώσεων, αλλά και ε, να δώσει στο Κοινοβούλιο την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αδιαφάνεια. Έχετε κάποια επιπλέον ερώτηση? Ναι, λέει η κυρία Τόγια, ευχαριστώ πολύ ε, για τις διευκρινήσεις. Ε, εγώ θα ήθελα από υποψήφια επίτροπο να μπορώ πολύ σύντομα να σας λέω, ε, να σας προσφωνώ επίτροπο αρμόδια για θέματα έρευνας, πολιτισμού κλπ. Αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά και για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια παρέμβασης, πιστεύω, όπως λέγατε και εσείς πιο πριν, να κατανοήσουμε τι γίνεται και με τα άλλα ταμεία τα οποία ασχολούνται με την καινοτομία και την έρευνα ε, εκτός Horizon αλλά με ισχυρή σύνδεση. Εσείς αναφερθήκατε και στο ε, Invest EU. Υπάρχουν ε, και υπάρχει το Digital Europe, υπάρχουν άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα κέντρα έρευνας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν κάποιοι κανόνες ε, και κάποιες κατάλληλες ε, ε, διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια ε, το έχουμε πει επανειλημμένα, οι συνέργειες δεν πρέπει να μένουν μονάχα κενό γράμμα, ε, αλλά όλοι κατανοούμε ότι ε, η πράξη είναι δύσκολη. Ναι, αναφέρθηκα ε, προηγουμένως και στο InvestEU, αλλά υπάρχει και το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Ε, όσον αφορά το Τίμινγκ, Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ε, κέντρο αριστείας οπωσδήποτε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να ε, βοηθήσει στη δημιουργία δομής που μετά το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο θα, θα μπορεί να χρηματοδοτήσει έτσι ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και οι υπηρεσίες μου και εγώ να δεσμευτούμε έτσι ώστε πριν από την υλοποίηση ε, των προγραμμάτων να έρθουμε, του το Horizon Europe δηλαδή, ε, να πάμε στις διάφορες χώρες, ε, να έρθουμε σε επαφή με τους υπεύθυνου, να μιλήσουμε, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ωραία, ωραίες συζητήσεις, καλή ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, αλλά δεν θα μας βοηθήσει εάν δεν βάλουμε και την πρακτική μέσα. Νομίζω πάντως ε, ότι ε, είναι πολύ σημαντική η πρόκληση. Ευχαριστούμε. Επόμενη μου κυρία Τζόνα Ντάουνινγκ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ για την ένταξη διαστάση του κλίματο σα πολιτική. Η έρευνα και νοτομία είναι βασικό σημείο για να φτάσουν μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2050. Κάτι που υποσχέθηκε η εκλεγμένη πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω τα στοιχεία του προπολογισμού για το 2020 του Ευρωπαϊκή Ενώσεω δείχνουν ότι ορίζοντα 2020 δεν θα πετύχει του στόχου αυτού για το κλίμα του 35%. Και ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε υπερεκτιμήσει όσον αφορά τη συνεισφορά του κλίματο στα πλαίσια του προγράμματο. Εμεί οι πράσινοι ανησυχούμε, διότι το, ο στόχο για το κλίμα το Horizon Europe θα τύχει της ίδιας μοίρας. Λοιπόν, πώς μεταφράζεται την αύξηση των φιλοδοξιών του 2050 στο ορίζοντα Ευρώπη με συγκεκριμένα μέτρα και οικονομικούς πόρους. Θα δεσμευτείτε να σταματήσει η χρηματοδότηση έρευνα και ανάπτυξη που είναι ει βάρο του κλίματο, κυρίω που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα δρομολογήσετε για να εξασφαλίσετε ότι ο ορίζον Ευρώπη πράγματι θα πετύχει του στόχου για δαπάνη για το κλίμα τουλάχιστον 35% και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σαν λογιστική άσκηση αυτό. Τι συγκεκριμένου μηχανισμού θα δημιουργήσετε σε περίπτωση ε, κενών και προβλημάτων και μη επίτευξη των στόχων και λήψεων χρημάτων. Κυρία Γκάμπρελ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ναι, καθορίσαμε το στόχο το 35% του προπολογισμού για το κλίμα. Τώρα πλέον είναι σαφές ότι τον ορίζοντα 2020 δεν θα αποτύχουμε, πετύχουμε το στόχο μας στο 30%. Αυτό που χρησιμοποιούμε για να προσμετρήσουμε αυτό το ποσοστό είναι ε, το ε, συγκεκριμένους δείκτες. Έχουμε ένα εργαλείο που έχουμε από τον ΟΣΑ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι κάθε πολιτική που με τον προπολογισμό άμεσα συμβάλλει σε στο στόχο το κλίμα θεωρείται ότι είναι στόχος 100%, δευτεροβάθμιο 40% και 0% παίρνει αν είναι κάτι άλλο. Έχω επίγνωση ότι ίσως δεν είναι τέλεια όλα αυτά τα μέτρα, είδαμε ότι είμαστε το 30% και το 30%, 35% δεν τα πετυχαίνουμε. Όμως για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την κατηγορία, αυτούς τους δείκτες του ρίου για να προσμετρήσουμε τις αποδόσεις. Αναμένω και κάποιες βελτιώσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν όλοι εκείνοι που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ούτως ώστε να το έχουν αυτό υπόψη όταν προετοιμάζουν τις διάφορες δράσεις να φροντίσουμε να έχουν περισσότερα ποιοτικά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε και την παρακολούθηση. Και εκεί θέσατε ένα θέμα ε, για το οποίο παραμένω ανοιχτή. Θέλω να ακούσω περισσότερες ιδέες. Για μας προφανώς είναι σημαντικό να δοθεί η συνέχεια. Προφανώς για μας είναι σημαντικό τη στιγμή που θα δούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί να μπορούμε να παρέμβουμε τάχιστα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται υπενθυμίζω ότι έχουμε μηχανισμό αξιολογήσεως και παρακολούθησης που εφαρμόζουμε κάθε χρόνο. Ίσα στα πλαίσια του κλίματος θα μπορούσαμε εδώ να τα καταφέρουμε καλύτερα. Το λέω σαφώς. Σήμερα είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Αν θέλουμε να πετύχουμε την κλιματική μετάβαση, αν θέλουμε να έχουμε αυτό το πράσινο σύμφωνο το ευρωπαϊκό, αυτό δεν θα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την έρευνα και την καινοτομία. Και γι' αυτό προφανώ θα υποστήριζα όλα αυτά τα προγράμματα που θα επιτρέψουν να μειώσουμε τι εκπομπές και να έχουμε επενδύσει ε, κατάλληλες και άλλες λύσεις που δεν γνωρίζουμε ακόμα και γι' αυτό έχουμε τα μέσα, όχι μόνο τον ορίζοντα Ευρώπη, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Έρευνας διαθέτουμε. Έχετε διευκρινιστική ερώτηση. Κυρία Ντάουτινγκ, οι περισσότερε συνεισφορά για το επίτευξη του στόχου για το κλίμα θα είναι από τα προγράμματα του ορίζοντα. Τι προγράμματα θα υλοποιήσετε για να αυξήσετε τα δύο κάτωθεν τμήματα για, τα, για την αξιολόγηση, για τα κριτήρια αξιολόγησης. Συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς θα εξασφαλίσετε ότι στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομία για κεφαλαιοβόρου τομεί, και δεν θα μένουν εκτός τα προγράμματα σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία, βιοτεχνολογία κλπ που εγγυούν, εγγυώνται ταχύτερη απόσβαση των επενδύσεων. Δηλαδή πώς θα είναι δυνατόν να μην περιθωριοποιούνται κάποιες τεχνολογίες που θα δίνουν σωστή λύση. Απάντηση, εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάποια επιλογή που δεν θα γίνεται σύμφωνα με κριτήρια στα οποία πιστεύουμε. Ε, υπάρχει μία λέξη, λύση, διαφάνεια. Θέλουμε να ξέρουμε πώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Καινοτομία επιλέγει τα προγράμματα θα πρέπει τακτικά να λαμβάνουμε πληροφορίε πώ γίνεται η επιλογή των λόγω προγραμμάτων. Θα ήθελα εδώ να τονίσω και κάτι άλλο, άλλα είδη μέσων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, κυρίω ψηφιακού τύπου. Την περσμένη εβδομάδα, στο Innovation και Research Day, ξεκινήσαμε μια νέα πλατφόρμα. Η κυρία Τόγια θα ενδιαφέρεται για αυτό, που αφορά τα αποτελέσματα του Horizon. Να μπορούμε να έχουμε βέλτιστε πληροφορίε όσον αφορά εκείνου που ετοιμάζουν τα προγράμματα, τι προϊόντα και τι αποτελέσματα πετυχαίνουν και οι χρήστες οι ενδεχόμενοι να μπορούν να ε, είναι πιο καλά πληροφορημένοι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει περιθώριο, μπορούμε να ισχύσουμε μέσω ψηφιακών μέσων περισσότερο τη διαφάνεια. Αυτή την ενιαία θηρίδα να την κάνουν πραγματική θηρίδα εισόδου όπου οι δικαιούχοι και οι νοησερχόμενοι θα μπορούν ε, εξακριβώς να επαληθεύουν τις διάφορες πληροφορίες και να ενημερώνονται. Ευχαριστώ. Χάνω Επιστροπής ε, πολιτισμού για το ID. Ευχαριστώ. Σαν μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, λέει ο κ. Ντάρε, εποφάσισε στο παντόχατο φυλάκιο που αφορά τον πολιτισμό, την εκπαίδευση νέους και αθλητισμό, είναι την καινοτομία και την νεολαία έχει εντάξει σε αυτό το ευρύτατο πλαίσιο. Το ίδιο έκανε η κυρία Ούρσουλα Βαντελάιεν και δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη πολιτισμού σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ποια οικονομικά μέσα θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των πολιτιστικό και δημιουργικό και για τη διαφύλαξη τη πολιτιστική κληρονομιά. Τι δράσει προτίθεται να θετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργηθούν δίκτυα πανεπιστημίων ευρωπαϊκών και κέντρων αριστεία, για την εκπαίδευση και για την επαγγελματική κατάρτιση. Τέλο, δεν, δεν τονίστηκε το σημαντικό το θέμα της αναπηρίας και του αθλητισμού και τη σχέση που έχει αθλητισμός με την αναπηρία. Τι οικονομικά μέσα αποτίθεται να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη, την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαμπριέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σας. Να τονίσω ότι υποστηρίζω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε ό,τι αφορά τον κλάδο του πολιτισμού, γιατί πιστεύω ότι εκεί πραγματικά μπορούμε να υπολογίζουμε στην δημιουργικότητα και στην καινοτομία. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Ό,τι αφορά καταρχά το Creative Europe και ό,τι υπάρχει ήδη σε ό,τι αφορά τα διατομιακά αυτά προγράμματα, σε ό,τι αφορά την δημιουργικότητα, τα εργαστήρια αυτά, Creative Innovation um, Laboratories, θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτή την πρόσβαση και υποστηρίζω λοιπόν τα προγράμματα αυτά και σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα στο ε, ορίζοντα Ευρώπη για να υπάρξει και μεγαλύτερη ορατότητα των διαφόρων αυτών παραδειγμάτων που υφίστανται σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Είμαστε στην αρχή του δρόμου και γι' αυτό λοιπόν για να μπορέσει να υπάρξει υλοποίηση αυτή του ωραίου αυτού οράματος, θα πρέπει να κοιτάξουμε 7 Νοεμβρίου τι γίνεται. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θα θέσω είναι η εξή. Έχετε ένα κοινό στρατηγικό όραμα ότι θα κινηθείτε προς την διακατεύθυνση. Ε, θέλουμε όλοι να έχουμε στρατηγικά προγράμματα κοινά, προγράμματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουν την κινητικότητα που θα επιτρέψουν η εκπαίδευση και η επικλιματική κατάρτιση να ληφθούν σωστά υπόψη αυτά τα θέματα θα τα υποστηρίξω, γιατί είναι σημαντικό λοιπόν ε, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα σήμερα. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις λοιπόν αυτές. Η έρευνα λοιπόν μπορεί να βοηθήσει πολύ να λάβουμε στην υπόψη τη διάσταση της έρευνας. Αν δεν θέλουμε να βρεθούμε σε πέντε χρόνια σε ένα χάσμα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα τα εκπαίδευση και τα προγράμματα ε, πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, είμαι πολύ ανοιχτή. Όπως σας είπα, είμαι υπέρ της αρχής της συμπερίληψης, ακόμα και για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να δημιουργηθούν ε, σχέσεις με, με ε, που θα πρέπει να δίνουν ελεύθερη πρόσβαση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ακριβώς αυτές τις νέες πρωτοβουλίες. Έχετε μία ερώτηση, κύριε Ταρέ. Είναι ερώτηση. Κοιτάξτε, Έκλεισε. Στον κόσμο της αναπηρίας χρειάζεται την Ευρώπη. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί από εμά. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και η κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού είναι κάτι εξαιρετικό. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση σε εσά, στην, ευαισθη... στην ευαισθησία σα, στο όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να, ρίξετε, να, έχετε, ρίξετε, να μην αποστρέψετε το όμορφο σα από αυτά τα άτομα. Κυρία, Κύριε Κάμπρελ, θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την έκκληση. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να πω το εξή. Το πρόγραμμα Europe for Culture είναι πολύ όμορφο. Μήπως να μπορέσουμε να σκεφτούμε το Europe for Sport από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι η κυρία Ντάτσε Μελπάρτε, που είναι συντονίστρια τη Επιτροπή ε, Πολιτισμού για το ECR. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ursula von der στην ατζέντα της για την Ευρώπη μιλά για την ε, θέση τον είπα σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ε, πόλο έλξης που αποτελεί για τα καλύτερα μυαλά. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η μάχη για τα καλύτερα μυαλά δεν αποτελεί μόνο μια εξωτερική πρόκληση, αλλά και ε, λόγω εσωτερικής τριβής και εσωτερικού ανταγωνισμού. Στη μάχη λοιπόν για αυτά τα καλύτερα μυαλά, το ανατολικό τμήμα της Ευρώπης φαίνεται να χάνει. Αυτή η μετανάστευση λοιπόν είναι αρνητική σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Brain drain, διαρροή εγκεφάλων, το αναφέρατε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Επηρεάζει πολύ σοβαρά το βιώσιμο μέλλον των κοινωνιών αυτών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ε, επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής αν δεν ανακοπεί αυτή η τάση. Ρωτώ λοιπόν, Πώς βλέπετε το σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ε, Εκπαίδευσης προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία σε ό,τι αφορά το σκέλος αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Καταρχάς, θα ήθελα να πω εν συντομία το εξής θα θέλαμε να ανανεωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Εδώ θέλω να κοιτάξουμε το θέμα του brain drain και το πώς μπορούμε να διατηρούμε τα καλύτερα μυαλά. Και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα βέλτιστα παραδείγματα. Και ο χώρος έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένας τέτοιος κλάδος Οι καλύτεροι ερευνητής θέλουν να παραμείνουν στην Ευρώπη. Αυτό που με ενδιαφέρει ακόμα πιο πολύ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας. Είμαστε ε, περήφανοι για τα βραβεία Νόμπελ και αυτό που κοιτάω είναι ότι ένας ε, ερευνητής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θέση απασχόλησης αλλά έξι άτομα. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται μια νέα α, κοινότητα ερευνητών. Έχουμε πάρα πολλούς διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και θα ήθελα να σας πω το εξής. Θα πρέπει στη συνέχεια να κοιτάξουμε και το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων. Αυτό αποτελεί μεγάλο θέμα σε πολλές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια διπλή βάση σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα Ευρώπη. Δεσμευτήκαμε προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίση τι δυνατότητε ε, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Marie Curie. Να δούμε τι δυνατότητε υπάρχουν για να δίνονται υποτροφίες για τα άτομα τα οποία θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους, γιατί υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα από πέρσι σε ό,τι αφορά την Γενική Διεύθυνση Έρευνας ε, για τα άτομα τα οποία έχουν κάνει έρευνα, έχουν πάρει χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020 για, που δεν έχουν λάβει μάλλον χρηματοδότηση, αλλά τους δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήταν εξαιρετικά τα προγράμματα τους και παράλληλα έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί οι ερευνητέ που κάνουν τέτοια προγράμματα. Είναι μεγάλο ο πόλο έλξη. Και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε και ένα θέμα πιο ευαίσθητο, του μισθού των ερευνητών. Έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε μία έρευνα για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Είμαι βέβαιη ότι αυτή η εξέλιξη θα μα δώσει πολλέ πληροφορίε για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε πιο γρήγορα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Έχετε κάποια συγκλονιστική ερώτηση, κυρία Μερμπαρντέ. Ναι, έχω μια ερώτηση σχετικά με την στρατηγική εξειδίκευση. Ποιο θα είναι ο ρόλος αυτή τη Smart Innovation Strategy στον σχεδιασμό της του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ε, οι στρατηγικές ε, εφιούς ε, εξειδίκευσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει πάρα πολλά και που βοηθάει και τις περιφέρειες να έχουν αυτήν την ευφυή στρατηγική εξειδίκευσης που μπορούν να μας επιτρέψουν περαιτέρω συνέργειες. Έδωσα και το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να επιτρέψει να δημιουργηθεί μία υποδομή ε, που αναφέρεται σε ένα άξονα που ήδη εμφανίζεται στην ε, στρατηγική εξειδικευσή και μετά ε, να έχει την δυνατότητα πρόσβασης στην χρηματοδότηση μέσω του Horizon Europe έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη γνωστοποίηση, μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των ε, περιφερειών. Ε, πραγματικά ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να έχουν γίνει ήδη αρκετά. Επίσης και η πρωτοβουλία περιφερειακής ανάπτυξης του είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Επόμενη Ομιλήτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Μέιντελ. Ε, κυρία Γκάμπριελ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσετε να οικοδομείτε στη σχέση αυτή και στο μέλλον. Ε, είπατε πολλά και ενδιαφέροντα στην ε, ε, εισαγωγή σας, μεταξύ των οποίων αναφερθήκατε εις τους μεγάλους αντιπάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία. Η ερώτησή μου είναι η εξής πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή έρευνα ε, θα ε, είναι ε, καλή για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, δηλαδή αυτές τις key enabling technologies. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάιντελ για την ερώτησή σας. Όπως το είπατε, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βασίζεται στην βιομηχανία της. Εάν θέλαμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε, να εξακολουθούμε να είμαστε μια Ευρώπη ε, που έχει την ικανότητα να ε, δίνει αποτελέσματα βάσει των υπεσχημένων στους ε, πολίτες θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, έχουμε αυτήν την τεχνολογία η οποία θα καθορίζει τα πρότυπα. Εάν δεν είμαστε εμείς και η δική μας τεχνολογία που θα καθορίζουμε τα πρότυπα, τότε ε, θα, ξεφύγουμε από τις ε, αρχές μας. Επαναλαμβάνω και κάνω αναφορά στην ε, κυβερνοασφάλεια, κάνω αναφορά επίσης εις την ε, τεχνητή νοημοσύνη στην οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες ε, προόδους. Επίσης ε, το, το θέμα του κοινού χώρου έρευνας αναφέρθηκε προηγουμένως στην τεχνητή νοημοσύνη ε, αλλά βεβαίως υπάρχει η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα, οι κβαντικές ε, αρχές, ε, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την ε, ισχύ της Ευρώπης, εκεί που η Ευρώπη μπορεί να έχει μια πραγματικά προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στον καθορισμό των προτύπων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε γιατί ο ορίζον ε, Ευρώπη ε, όντως βρίσκεται στο, διαφαίνεται στον ορίζοντα αλλά υπάρχουν ε, και τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινού συμφέροντος. Το κάναμε για τα Photonics, θα το συνεχίσουμε και με άλλους τομείς. Επομένως, για μία ακόμα φορά εγώ λέω ότι αν θέλουμε πραγματικά να καταφέρουμε να επιτύχουμε την αυτονομία, εάν θέλουμε να μην χάσουμε το νέο κύμα ε, ε, ε, επένδυσης στην έρευνα, πραγματικά τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τις επενδύσεις. Τώρα είναι η ώρα τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε μία επερώτηση. Κυρία Μέιντελ, ναι. Ε, γνωρίζετε ότι η στρατηγική αυτονομία ε, αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και για αυτά τα οποία ε, καλά τα καταφέρνουν στο Horizon Europe και για τις άλλες χώρες που δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Συνέργειες μεταξύ του προγράμματος ε, Horizon και άλλες νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες καθώς επίσης και άλλα ταμεία έτσι ώστε να διευρυνθούν τα εργαλεία τα οποία μπορούν και θα μπορέσουν και στο μέλλον να φέρουν κοντά την ερευνητική κοινότητα και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι, καταλαβαίνω ε, τι λέτε. Ε, στην ουσία ήδη είμαστε σε θέση να μιλάμε ε, για το Περιφερειακό Ταμείο, για το Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Τα ανέφερα και προηγουμένως άλλωστε και τα ανέφερα και σε σχέση με τα προγράμματα αριστείας. Ε, αυτά τα προγράμματα αριστείας έχουν, ε, δίνουν την δυνατότητα γρηγορότερης πρόσβασης ε, στα κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια και το αναφέρατε κι εσείς, τα κράτη δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο σημείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει η προσπάθεια και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για πρώτη φορά ε, βλέπουμε ε, μέτρα για teaming ε, και παρόμοια προγράμματα τα οποία φτάνουν σε ένα τμήμα της τάξης του 3,3% από του, γενικού προϋπολογισμού. Θέλω να πω ότι μπορούν να υπάρξουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα, τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα πάντα με διαφάνεια έτσι ώστε να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Σα υπενθυμίσω παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο που είναι στη διάθεσή σα διότι τελειώνει ο χρόνος μας. Η Βασιλιάψ από την Επιτροπή Ήτρε και από τη Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, καλωσορίζω τους τέσσερις τομείς δράσης, τις τέσσερις άξονες δράσης που αναλαμβάνετε για να καλύψετε τα κενό καινοτομία εκείνων που λυγούνται, εκείνων που έχουν μείνει πίσω και να μειωθεί και η φυγή εγκεφάλων. Ανησυχητικό το κενό στην έρευνα και τεχνολογία. Είχε μείνει πίσω η Ευρώπη. Έχουμε διάλογο στα πλαίσια του ορίζοντα, αλλά οι συνέργειες εξαιρούνται με άλλα προγράμματα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το ιδεώδες σύστημα συνεργειών του Horizon Europe με άλλα ερευνητικά προγράμματα για να καλυφθεί το κενό στην έρευνα και καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όπως είπατε, αυτό που είναι σημαντικό για μένα στο πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι να δούμε πώς τα νέα κονδύλια για την διεύρυνση του widening θα δώσει λύσεις όσον αφορά το χάσμα που δημιουργείται. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινή προσέγγιση αν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις, όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γι' αυτό θα υποστήριζα πραγματικά τα νέα μέσα, τα νέα εργαλεία, κυρίως τη δυνατότητα να μπει κανείς σε ένα δίκτυο, να μπορεί να μπει σε διάφορα κονσόρτσια και θα πρέπει να δούμε πόσα κράτη-μέλη χρησιμοποιήσουν τις ε, δυνατότητες που δίνουν τα άλλα ταμεία οι άλλοι πόροι για να δημιουργηθούν περισσότερες συνεργασίες. Εκεί προσπαθούμε κάπως να προδικάσουμε τη διαδικασία. Πριν ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις συνέργειες, υπέχουμε καθήκον να έχουμε σαφέστατο ορισμό των συνεργασιών αυτών να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τα εργαλεία που διαθέτουμε και πιστέψτε με αυτό ακόμα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό εγώ θα προσπαθήσω να πείσω τους άλλους συναδέλφους επιτρόπους, να τους πείσω πόσο σημαντικό είναι σε κάθε μία από τις αντίστοιχες πολιτικές τους είναι να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την έρευνα και καινοτομία και να λάβουν υπόψη την αξία τους και να μπορέσουμε να έχουμε αυτού του είδους τα εργαλεία. Δεν είναι μόνο το Ταμείο της Συνοχής, δεν είναι μόνο το Digital Europe, δεν είναι μόνο το Invest EU. Όλα αυτά θα πρέπει να αποκτήσουν ε, σάρκα και οστά. Θα είμαι πολύ προσεκτική γι' αυτό. Βλέποντας το κείμενο το νομικό του πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, οι συνέργειες εντοπίζονται με 20 άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κινητικότητα μέχρι κοινωνικό ταμείο, περνώντας πολλούς άλλους τομείς. Αυτό που θα πρότεινα να κάνουμε τώρα θα ήταν το εξής πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για την σημασία των επενδύσεων για καινοτομία, γίνεται η συζήτηση, θα πρέπει να επασπιστούμε τα ποσά που προβλέπονται, θα πρέπει να έχουμε το χρόνο, να έχουμε ένα χρόνο στη διάθεσή μας, να δώσουμε προσανατολισμό σε επενδύσεις. Τώρα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για σωστό προβληματισμό. Βασικά σημεία εντοπίστηκαν, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που προσήξαν την, προσοχή μου. Ο στατηγικός σχεδιασμός θα αποτελέσει ένα καλό μέσο για να πετύχουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γέψη, έχετε μια διευκρινιστική ερώτηση. Ναι, ναι. Εξής ερώτηση. Πώς θα πείσετε όχι μόνο τους συναδέλφους επιτρόπους, αλλά και τα κράτη-μέλη να διοχετεύσουν περισσότερα χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία για υποδομές, για έρευνα και ανάπτυξη και για να διευκολύνουν την μεταρρύθμιση που απαιτείται για την έρευνα και την καινοτομία και τα συστήματα πολλών χωρών σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση με τα κράτη-μέλη. Μία προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί αναχώρα. Οι ανάγκες δεν είναι ίδιες, οι υποδομές δεν είναι ίδιες. Κάποιες Καλές πρακτικές υπάρχουν σε κάποιες χώρες, σε άλλες δεν υπάρχουν. Θέλω να έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, να δούμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία. Όπω σα είπα, έχουμε κάποια καλά παραδείγματα. Τέσσερι χώρε πέτυχαν το στόχο του 3%. Άλλε δεν πέτυχαν το στόχο, αλλά ανάμεσα σε αυτέ υπάρχουν και άλλε. Εγώ, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία, τέσσερι χώρε που έκαναν πολλέ προσπάθειε τα τελευταία χρόνια παρόλο που ε, υπολείπονται του στόχου. Αυτό που ήταν σημαντικό αυτή τη στιγμή θα ήταν σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Να μην τους λέμε ότι υπάρχουν συνέργειες, να πούμε πώς στα πλαίσια τα δικά τους, συγκεκριμένη τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές, τις υποδομές, την πρόοδό του, την τεχνολογία του, τι επενδύσει που υπάρχουν για έρευνα και ανάπτυξη, να του δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα μέσα ε, αυτή την εμπειρία έχω αποκομίσει. Πολλές φορές άκουσα αυτή την ανάγκη να μην μένουμε μόνο σε γενικόλογες ε, δηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη μεγήτρια, η κυρία Κλέρ Φόξ από την Ήτρα και την Επιτροπή Πολιτισμού από τους μη Γραμμένους Κυρία Γκάμπριελε, ένας βασικός τομέας στην έρευνα και την ανάπτυξη και στα πανεπιστήμια είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία που απειλείται σε πολλά κράτη και διεθνώ. Θα ήθελα μια επιβεβαίωση από πλευρά σα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τα προηγούμενα χαρτοφυλάκια σα, ότι η έρευνα που χρειάζεται για την παραπάνω πρόσβαση στις ε, πληροφορίες online για παράδειγμα, αλλά παρόλα αυτά η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει να τεθούν οι παράμετροι για το να δούμε τι περιεχόμενο παραμείνει, online. Υπάρχει λοιπόν μία αντίθεση μεταξύ της ε, περιορισμού της ελευθερίας της λόγου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Είναι αρκετά περιορισμένη ο ορισμός σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΕΠΑ κτλ. σε ό,τι αφορά την εφαρμοσιμότητα. Και υπάρχει πιο πολιτικό σκέλος σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω της εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι όλα αυτά απειλούν την ακαδημαϊκή ελευθερία και απειλούν την έρευνα σε ό,τι αφορά για τη γνώση. Για τη γνώση. Έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού. Νομίζω ότι με κάθε ε, δύναμη θα προσπιστώ την ακαδηματική ελευθερία προκειμένου η έρευνα να καθοδηγείται από την περιέργεια και να μπορεί να υπάρχει. Πώς είμαστε να γνωρίζουμε παραδείγματα εφευρέσεων που προέκυψαν χάρη στην έρευνα που όταν παρουσιάστηκαν δεν γνωρίστηκε η σημασία τους. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνω ιδιαίτερως ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία μεταξύ της έρευνας, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Και εδώ λοιπόν υποστηρίζω την ευρωπαϊκή έρευνα για να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, τα σύνορα στην έρευνα, αλλά ότι σήμερα πιο πολύ παραποτέ μαζί με τους πολίτες θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο και τη διαφάνεια για να υπάρξουν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις, την αλλαγή του κλίματος, την ε, ψηφιακή μετάβαση και νομίζω ότι όλοι θέτουν ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά και τη βιομηχανική πολιτική. Αναφερθήκατε και σε ένα άλλο στοιχείο, στο θέμα της ανοιχτής επιστήμης. Αυτό αποτελεί ένα θέμα που το έχω μέσα στην καρδιά μου και θα εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί σήμερα πιο πολύ παραποτέ έχουμε ανάγκη να μπορούν οι ερευνητές να μοιραστούν τα αποτελέσματα της ερευνά τους με άλλους επιστήμονες και να μπορέσουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των άλλων. Οι δημοσιεύσεις λοιπόν που χρηματοδοτούνται από τον οριζόντα Ευρώπη θα πρέπει να δημοσιεύονται άμεσα, να γίνονται σεβαστές φυσικά κάποιε αρχέ. Όσο πιο ελεύθερη γίνεται και όσο πιο κλειστή ε, επιτάσσει η ανάγκη προκειμένου να έχουμε και τα θέματα δεδομένων τα οποία να χρησιμοποιούνται και να είναι ποιοτικά. Και σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα μπροστά μα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το πλαίσιο τη έρευνα. Πώ μπορούμε να ενθαρρύνουμε του ερευνητέ εκείνου που υποστηρίζουν την ανοιχτή επιστήμη αυτή την ελεύθερη πρόσβαση, γιατί καταβάλουν προσπάθειες τις οποίες άλλοι δεν τις καταβάλουν. Συμφωνώ ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να ασχοληθούμε για να είμαστε ισχυροί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε τη θέση μας μέσα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάποια συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Φόξ. Μάλιστα, ναι. Αυτό πραγματικά με καθεσυγάζει. Αλλά νομίζω ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συχνά αναμειγνύονται στα πανεπιστήμια. Και όταν υπάρχει ένα τέτοιο όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ξανακάνουμε το ίδιο. Και παρά την διαβεβαίωση που μου δίνεται σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε από την επιστήμη. Εγώ είμαι νευρική και αναρωτιέμαι επίση. πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε πιο σαφώς ε, τα πανεπιστήμια για τη γνώση καθεαυτή και την εκπαίδευση εκατομμυρίων ανθρώπων σε κρατη που δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, μιλώντας με κάποιους νεαρούς μηχανικούς στο βυτικό τμήμα της Βρετανίας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν μιλάμε για την διαρροή εγκεφάλων, συχνά μιλάμε για τα πανεπιστήμια, ενώ στην ουσία πολλά μεγάλα μυαλά είναι μαθητευόμενοι ε, άνθρωποι με δεξιότητες νέοι που συχνά τους ξεχνάμε στο πλαίσιο αυτό. Πώς μπορούμε λοιπόν και αυτούς να τους αθαρρύνουμε. Δεν μιλάμε μόνο για τους πανεπιστημιακούς φοιτητές. Το μήνυμά μου είναι απολύτως σαφές. Βεβαίως ε, δεν θέλουμε να κλειστούμε ε, είτε στα, στους τέσσερις τείχους ε, μιας, ενός σχολείου, ενός πανεπιστημίου. Η διαχωρισμοί δεν υπάρχουν όσον αφορά την ηλικία, την κατάρτιση κτλ. Εγώ θέλω να στείλω ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα γιατί αυτό είναι και ο στόχος του προγράμματος Erasmus Plus Θέλουμε μεγαλύτερο άνοιγμα όσον αφορά ε, τα εργαλεία που έχουμε. Ε, ε, σκέφτομαι άμεσα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία. Εκεί πραγματικά δίνονται νέες ικανότητες, γιατί ξέρετε δεν είναι δεδομένη ε, μια ε, παραδοσιακή κλασική διαδρομή ε, για όλους και εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή θα έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν υπόψη τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια το θέμα αυτό και με μια τελευταία λέξη στην ακαδημαϊκή ελευθερία για την ακαδημαϊκή ελευθερία πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ πιστεύω σε αυτήν και μαζί με την ελευθερία στην έρευνα αποτελεί αποτελεί μία από τις αρχές μας. Έχουμε τον χάρτα, την χάρτα για τα πανεπιστήμια και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου έτσι ώστε όλες αυτές οι αρχές να γίνουν σεβαστές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζούλι Ward από την Επιτροπή ΚΑΛΤ ε, για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ε, προβληματιζόμαστε ε, με τις ε, ε, επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι στην εκάλυψη των αρχών τους και επίσης όσον αφορά τα fake news που δυναμητίζουν, υπονομεύουν την δημοκρατία μας. Ε, πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκάμπριελ, για τις ερωτήσεις σας, διότι θίγεται ε, ζητήματα θεμελιώδους ε, σημασίας. μίλησαν προηγουμένως για την ε, ακαδημαϊκή ελευθερία, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και την καλλιτεχνική ελευθερία. Εγώ με ιδιαίτερη προσοχή θα αντιμετωπίζω και το θέμα αυτό. Νομίζω ότι και με την εξέλιξη του ψηφιακού κόσμου, αυτού του νέου ψηφιακού κόσμου, θα πρέπει ε, να σταθούμε και να μελετήσουμε τις νέες προκλήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε πλέον προσήκοντα εργαλεία πιο κατάλληλα εργασία. Ε, πρέπει ε, να το κάνουμε και το κάνουμε ήδη για την καλλιτεχνική ελευθερία. Θα διοργανωθεί σχετική ημερίδα την, τον επόμενο μήνα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές τις οποίες ε, όλοι σεβόμαστε και μας είναι ιδιαίτερος προσφυλής όσον αφορά την παραπληροφόρηση, της ψευδής ειδήσει fake news. Εδώ θίξατε ένα θέμα το οποίο πραγματικά βρίσκεται στην καρδιά μου. Υπάρχει αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην διαφάνεια, στην υπευθυνότητα, την ελευθερία έκφρασης ε, και την ελευθερία στη σωστή πληροφόρηση. Ήδη υπάρχει και μία πρωτοβουλία την οποία έχω υποστηρίξει. Είναι το Safer Internet for EU. Ε, βλέποντας ε, το σχέδιο ψηφιακής εκπαίδευσης, οι δύο πρωτοβουλίες μεταξύ των τριών πιο επιτυχημένων είναι το Codic και το Safer Internet for EU. Η εκστρατεία για το ε, ασφαλέστερο διαδίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ήδη καρπούς. Έχω πάει σε πάρα πολλά σχολεία και κατάλαβα ότι τα παιδιά θέλουν να γνωρίζουν και να έχουν δυνατότητα ε, πρόσβασης. Κανείς δεν θέλει να τους υποχρεώσει να διαβάσουν κάτι, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε οπωσδήποτε τα εργαλεία έτσι ώστε να έχουν την επιλογή, να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μετά από σωστή αντικειμενική κριτική σκέψη. Αυτά τα εργαλεία θέλουμε να τους δώσουμε. Όσον αφορά ε, το πρόγραμμα της ε, ε, προώθησης το, της παραπληροφόρησης εγώ θα ήθελα πιο πολύ να δούμε το θέμα από την άλλη πλευρά δηλαδή να προωθήσουμε προγράμματα media literacy αλφαβητισμού ή ενημέρωση όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Ε, επερώτηση, κυρία Ward, ναι. Μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τρίτες χώρες και για γειτονικέ ε, χώρες. Ποιος είναι ο ρόλος ε, των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων ε, γιατί νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε ε, και ένα πολύ, καλό, ένα πολύ καλό πεδίο συνεργασίας της Επιτροπής Πολιτισμού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες το θέμα του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τα ε, Βαλκάνια. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ε, την πολιτιστική στρατηγική στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. η πολιτιστική διπλωματία, λέει η κυρία Γκάμπριελ, είναι ε, μία μορφή ήπιας ε, διπλωματίας, ε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα μέσα της hard, της σκληρής διπλωματίας σκοντάφτουν και εκεί πραγματικά μπορεί η ήπια διπλωματία να παίξει καλό ρόλο. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, γιατί είναι χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρώπης και είναι χώρες οι οποίες θέλουν σήμερα να δουν την συγκεκριμένη μας υποστήριξη ε, και όσον αφορά το roaming βέβαια, αλλά και όσον αφορά ε, την ε, Δημιουργική Ευρώπη, Creative ε, Europe ε, και πραγματικά στην Σερβία είχα ένα παράδειγμα ανθρώπου που είδε τα μάτια του να λαμπυρίζουν όταν, τους, όταν του μίλησα για αυτήν την Creative Europe. Μιλάμε ε, για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι τις εγκαταλείπουν τις χώρες αυτές οι νέοι. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στις χώρες αυτές νέες προοπτικές και επομένως η δημιουργική βιομηχανία, ε, ε, η δημιουργία γενικότερα είναι κάτι ιδιαίτερο προσφυλές σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίες, για τις τελευταίες εξερωτήσεις δίνω ξανά την Προεδρία στη συνάδελφο την κυρία Βαλάν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Αντάμοφ από το ΕΛΚ, Επιτροπή Πολιτισμού. Въпросът ми е свързан с изравняването на възможностите между източна и... Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω για τι ευκαιρίε μεταξύ Ανατολική και δυτική Ευρώπη όσον αφορά το Horizon, το Creative Europe. Όσον αφορά το Horizon Europe, πολλά κράτη-μέλη έχουν χαμηλό ποσοστό εγκεκριμένων προγραμμάτων όπως η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ουγγαρία και άλλοι. Πώς θα προωθήσετε αυτό το πρόγραμμα να καλύπτει όλη την Ευρώπη, να εξασφαλίσουμε ότι η συμμετοχή των ανατολικών και των δυτικών κρατών θα υπάρξει δυνατότητα τεχνικής αρρωγής όσον αφορά το Creative Europe. Αυτό το πρόγραμμα τώρα ελέγχεται από διάφορους επιτρόπους και διάφορους γενικούς διευθυντής. Το υποπρόγραμμα ε, Media ε, υπό την υποπτήρια άλλου. Ε, πώς θα συντονίσετε το έργο μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Πώ θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Θα εξασφαλίσετε ότι αυτό το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί επαρκώ, ούτω ώστε να προωθήσει περισσότερο τον πολιτισμό και πρωτοβουλίε δημιουργικέ από όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάμοφ, για την ερώτησή σα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το ορίζον Ευρώπη. Το μήνυμα ακούστηκε σαφώς σήμερα. Το θέμα του widening σημαντικό, διεύρυνση. Είμαστε υπερήφανοι τώρα για το 3,3% του προπολογισμού που θα δοθεί για αυτό το σκοπό. Αυτό που θα με ενδιέφερε θα ήταν πραγματικά να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες να συμμετέχουν. Διότι όταν δούμε το ποσοστό συμμετοχής τη ε, της Ευρωπαϊκής των 13, 5,06% φέτος. Πέρσι ήταν 4,8% δείχνει ότι όταν έχουμε περισσότερα προγράμματα όπως η αδελφοποίηση για την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, teaming, ομαδοποίηση για τα κέντρα αριστείας, το SHARE, Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, όταν οι διάφοροι επιφανείς ερευνητές μπορούν να προχωρήσουν. Ε, προωθείται η έρευνα. Μετά θέτε ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 να έχουν περισσότερη ενίσχυση τεχνική. Πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα ε, και μέσα για τεχνική αρρωγή. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα επιτυχιών. Policy Support Facility είναι ένα μέσο διευκόλυνσης πολιτικών. Μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες με συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά αυτό μπορεί να έχει διαφορετική μορφή αυτή η βοήθεια. Μπορούμε να βοηθήσουμε μια χώρα συγκεκριμένη. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την αλόγω χώρα για συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορούμε να πειραματιστούμε ή ακόμα μπορούμε να έχουμε βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις που ε, εφαρμόζει σε άλλη χώρα και να ενημερώσουμε τη χώρα που βοηθάμε. Επίσης μπορούμε να δώσουμε χρήματα από τη τα ταμεία. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Υπάρχει μια σειρά εργαλείων αυτό που είναι σημαντικό είναι να τα γνωστοποιήσουμε, τόσο ώστε οι χώρες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά. θα περάσω το μήνυμα για αυτό το τμήμα της Ευρώπης που αναφέρατε και να το μάθει και αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Κύριε Αντάμοφ. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Αντάμοφ. Κοιτάξτε, στο χαρτοφυλάκιό σας θα έχετε την πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή έρευνα και την παιδεία και το σχετικό χώρο. Ο ευρωπαϊκός, ευρωπαϊκός χώρος για την παιδεία θα πρέπει να κινηθεί για την αναγνώριση διπλωμάτων. Πώς είναι αυτό δυνατόν αν όλοι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. Απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Παιδεία, Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης. Στόχος που έχουμε θέσει χρονικά είναι το 2025 για την υλοποίηση των στόχων μας. Για την ώρα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Όπως είπατε, ο ίδιος είναι θέμα που αφορά και τις εξουσίες των κρατών μελών. Πρέπει να δούμε τι προστιθέμενη αξία δίνει η ευρωπαϊκή συνεργασία, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλώντας τώρα για τον ευρωπαϊκό χώρο παιδείας, Ίσως εκεί θα πρέπει να βασιστούμε στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για να μπορεί να υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων. Όπως είπα, στόχο έχουμε θέσει το 2025. Υπάρχει κάτι άλλο. Συμφωνώ. Πράγματι θα έπρεπε να έχουμε Ευρωπαϊκή Κάρτα Φοιτητών μέχρι το 2021. Αυτή η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα θα επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα όταν είναι στο εξωτερικό. Δεν θα αντικαθιστά την εθνική όμως, αλλά αυτή είναι άλλη μια ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μίχελσα από την ΚΟΕ και την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. την κυρία Επίτροπε, ο Έλληνας ε, συναδελφός μου Αλέξης Γεωργούλης σε μια ανοιχτή επιστολή Προ την κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι χωρί πολιτισμό η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα ήταν ε, ασύλληπτη. Εσεί μιλήσατε για την πολιτισμό ως DNA της Ευρώπης. Θα ήθελα μία ξεκάθαρη απάντηση από πλευρά σας. Δεν πιστεύετε ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρος ε, στα, στη χρηματοδότηση, όχι μόνο στις περιγραφές και μία ερώτηση που σας είχα κάνει και το 2017, δεν την είχατε απαντήσει τότε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, συντακτών ε, και όλα αυτά τα ανοιχτά, εκρεμή ζητήματα, σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικών τα πνευματικά δικαιώματα. Πώς θα, τα καλύψετε, τι θα κάνετε με τα μουσεία, τι θα κάνετε με την ε, πρόσβαση online και offline. Πώς θα τα εξασφαλίσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κάπριελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξεκινήσω από την οδηγία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Ναι, κάναμε εξαιρέσει για την έρευνα, την εκπαίδευση, για τις βιβλιοθήκες, την πολιτισμική κληρονομιά. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο κείμενο. Αυτό που θα ήθελα τώρα είναι να συνεχίσουμε να ακολουθούμε την διαδικασία από κοντά για να δούμε πώς θα γίνει η υλοποίηση, η εφαρμογή. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε και άλλη μια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το κείμενο το πετύχαμε, το οποίο είναι πολύ σωστό. Χαίρομαι. Προφανώς θα πρέπει να δω πώς θα γίνει η υλοποίηση, η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Θα καταβάλω προσπάθειες για να ε, ενημερώσω ε, αυτούς που θα ωφεληθούν από τις εξαιρέσεις αυτές. Να αναφερθούμε τώρα στη συνέχεια στον πολιτισμό. Πίστευα πραγματικά ότι τα τελευταία χρόνια στο περιβάλλον ε, του πολιτισμού, οι συγγραφείς, οι δημιουργοί έχουν νιώσει πόσο έχουμε δεσμευτεί. Η επιστολή ε, αποστολής μου δεν κάλυψε με εξαιρετικό τρόπο όλα τα στοιχεία, αλλά ήμουν σαφέστατη ότι ο πολιτισμός για, μένα θα αποτελέσει πάντα ένα θέμα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου, γιατί σήμερα ο πολιτισμός, όπως είπατε, είναι η ευκαιρία που έχουμε για να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο συμπεριληπτική, πιο καινοτόμα. Μια Ευρώπη πολύ απλά η οποία θα λάβει πιο πολύ υπόψη την ποικιλομορφία προκειμένου να προωθήσει ε, μια ποικιλία ιδέων και καινοτομιών που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και θα μπορέσουμε να τα κοιτάξουμε όλα αυτά με μεγαλύτερη ακρίβεια και γι' αυτό ήμουν ξεκάθαρη. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την εθνική κληρονομιά. Θα ήθελα και θα εργαστώ προκειμένου ο πολιτισμός να παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, προκειμένου να έχουμε το ευρωπαϊκό πολιτισμικό κλειδοδότημα, το οποίο πλέον θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θα υποστηρίξω λοιπόν όλες αυτές τις ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Μιχέλση για μια διευκρινιστική ερώτηση. Ναι, αλλά παρόλα αυτά αυτό λείπει από την αποστολή σας. Η συνάδελφος Κάμερ ε, μίλησε για την οδηγία για τα πτυακοστικά μέσα. Θα ήθελα να ε, γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, κοιτώντα τα θέματα ευθύνη των συγγραφέων, των δημιουργών σε ό,τι αφορά τι πλατφόρμες ε, για το video sharing. Αν όλα αυτά θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε από πολιτικό τρόπο, με πολιτικό τρόπο, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την ε, οδηγία για το e-commerce, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κυρία Γκαμπριέλ. Θα είμαι σύντομη. Ναι, πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες μας για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ψηφιακή μετάβαση και να αποκριθούμε στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φίστο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, από την ΙΤΡΕΜ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Γκάμπριελ, για την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος Ορίζοντας 2020, Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλο χάσμα μεταξύ των παλαιών και των καινούργιων κρατών μέλων σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προγραμμάτων και τη χρηματοδότηση. Το παράδειγμα αυτό έχει αναφερθεί πολλάκις τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα έχουν μία βασική, ένα βασικό πρόβλημα, δύσκολους όρους εφαρμογής και αυτό δεν δίνει οι ίδιες ευκαιρίες στα πιο έμπειρα και στα λιγότερο έμπειρα κράτη-μέλη. Πώς θα αναρμονίσετε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου ο Ορίζον Ευρώπης να καταστεί ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει πιο πολλές χώρες. Έχετε υπόψη σας συγκεκριμένα μέτρα για να υποστηρίξετε την επιστημονική κοινότητα στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης θα ξεκινήσετε μαζί με τα Υπουργεία των Κρατών Μελών νομοθετικές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί το χάσμα το μισθολογικό σε ό,τι αφορά τους ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χριστόφ. Θα ήθελα να απαντήσω λακωνικά. Διεύρυνση του πεδίου κάλυψης Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αποδοτικά όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα. Είπατε μία λέξη που είναι πολύ σημαντική. Απλούστευση. Απλούστευση ισχύει για ένα κομμάτι των διαδικασιών που αφορούν τον ορίζοντα 2020. Θα προχωρήσουμε και πιο πέρα. Διότι απλούστευση είναι το πνεύμα που στηρίζει τα νέα προγράμματα του Ευρώπη, Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τρεις πυλώνες με σαφέστατη λογική παρέμβαση. Σε κάθε πυλώνα, από την έρευνα στην καινοτομία, έχουμε σαφή περιγραφή του μηχανισμού που έχει σαν στόχο την απλούστευση. Και αυτός ο μηχανισμός θα στηρίζει και θα καθορίζει τα προγράμματα και τη συμμετοχή. Να προσέξουμε ιδιαίτερα την απλούστευση των διαδικασιών. Γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται όλοι. Θέλουμε να έχουμε ένα είδος εγγράφου, εντύπου όσον αφορά τις αιτήσει για τη συμμετοχή. Να ζητάμε λιγότερες πληροφορίες από τους μελλοντικούς δικαιούχους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερα προγράμματα που θα εντάσσονται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης και πρέπει να έρθουμε στο θέμα των πληρωμών των μισθών, των ερευνητών. Όταν πληρώνονται για ένα πρόγραμμα, ο μισθός τους βασίζεται επί των επιπέδων των μισθών σε κάθε χώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα άμεση παρέμβασης. Όμως θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει θα παρακολουθήσουμε ποια είναι η εξέλιξη των μισθών των ερευνητών στην Ευρώπη. Θα γίνει μελέτη, θα δούμε πού υπάρχουν οι μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις αμοιβέ, τους μισθούς των ερευνητών, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας και έτσι θα δούμε κάποιες διεξόδους ε, για την εξέβρεση λύσεων. Όπως ξέρετε τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που μπορούν να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς μπορούμε μόνο να βοηθήσουμε. Κύριε Χριστόφ, έχετε διευκρινιστική ερώτηση. Σύντομα παρακαλώ ο κύριος Κριστόφ. Έχετε συγκεκριμένα μέτρα που μπορείτε να αναφέρετε για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής έρευνας για να σταματήσει η φυγή των εγκεφάλων, το brain drain. Είπατε ότι δεν υπάρχουν πολύ συχνά τα κατάλληλα χρήματα. Δεν υπάρχει δεν θέλουμε να υπάρχει διακίνηση μεταξύ ευρωπαϊκών. Θέλουμε διακίνηση των σπουδαστών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην φεύγουν και να πηγαίνουν ε, στο εξωτερικό στη ΗΠΑ. Περισσότεροι Βούλγαροι σπουδάζουν στο εξωτερικό από ότι στη Βουλγαρία. Και τελικά θα δημιουργηθούν σε κάποια μέρη της Υπήρου μας κάποια σπουδαστικά γκέτο με αυτόν τον τρόπο. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ το έχω ήδη ξαναπεί θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να δούμε τι θα συμβεί με τις υποτροφίες Μαρή Λοντόφσκα Κιουρί. Ε, γιατί θέλουμε να δούμε ε, κατά πόσον μπορούν να, ε, να χρησιμοποιηθούν αυτές ε, οι υποτροφίες και μετά να επιστρέψει στην χώρα προέλευσης ο ενδιαφερόμενος. Ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιες υποτροφίες που θα δίνουν την δυνατότητα στους επιστήμονες αφού θα έχουν εργαστεί στο εξωτερικό να επιστρέψουν στις χώρες τους. Οπωσδήποτε θα πρέπει να παρακολουθούμε τις, εξελίξεις, τις εξελίξεις, συγγνώμη, διότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όσον αφορά τις διαδικασίες και ε, επομένως ε, θα πρέπει να δούμε ακόμα και από ιεραρχικής απόψεως και από άποψη διαφάνειας πώς έχουν τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, το είπα και το ξαναλέω, ε, να υπάρχει και ένα ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβών μισθών. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μέχρι το 2024 τα ευρωπαϊκά αυτά πανεπιστήμια. Η Αντιπρόεδρος... Ε, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού. Όταν η ακροδεξιά προχωράει και ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η φοβία των ε, ΛΟΑΔ, ο αντισημιτισμός και άλλα κακά α, κορυφώνονται. Πώς σκοπεύετε να, να καταπολεμήσετε αυτά τα φαινόμενα με αποτελεσματικό τρόπο. Το Erasmus Plus είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το διαπολιτισμικό διάλογο και την προώθηση του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής ε, σλόγγανα ε, ενωμένη στην πολυμορφία. Δεσμεύεστε να έχετε στόχου σε ό,τι αφορά τα άτομα με περιορισμένες ε, ευκαιρίες. Πώς θα κάνετε λοιπόν το Εράσμος πιο προσβάσιμο και πιο συμπεριληπτικό. Να σας υπενθυμίσω, η εκπαίδευση δεν είναι ακόμα προσβάσιμη σε όλους στην κοινωνία μας. Ε, δεν ε, αντιμετωπίζονται όλοι με τους ίδιους όρους. 80% των ατόμων με προέλευση Ρωμά στη Γερμανία δεν έχουν σωστή πρόσβαση στην εκπαίδευση και το μέλλον τους είναι προδιαγραμμένο. Βασικός ε, λόγος είναι ο ρατσισμός. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση, πώς μπορεί να προετοιμάσει κανείς τους νέους, να τους δώσει εφόδια για να μην πέσουν σε αυτήν την παγίδα. Βεβαίως το πρόγραμμα Εράσμους παραμένει ένα καλό πρόγραμμα ε, για το θέμα αυτό, ακόμα και τώρα έχουμε αυτά τα ε, σχέδια τα οποία επιτρέπουν στους νέους ε, να δουλέψουν με τρόπο ώστε η ριζοσπαστικοποίηση ε, να μην είναι στην ημερήσια διάταξη. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι μια κατάσταση σαφής όλων των projects, να δούμε ποιο είναι αυτό που λειτουργεί, ποια είναι αυτό που δεν λειτουργεί, γιατί διαβάζω τα χιλιάδες προγράμματα Erasmus και κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα είναι μοναδικό. Όμως πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε να μπορούμε να εξάγουμε δύο ε, δάγματα τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη κατάσταση. Η ριζοσπαστικοποίηση δεν γίνεται μονάχα στο φυσικό κόσμο. Πιστεύω ότι κυρίως γίνεται ε, στον επιγραμμικό κόσμο. Γι' αυτό ε, έχω πραγματικά υποστηρίξει την εκστρατεία για το ασφαλέστερο διαδίκτυο και για ε, την προετοιμασία των νέων ε, για την χρήση του διαδικτύου και πώς τα δικά του στοιχεία χρησιμοποιούνται έτσι ώστε πολύ ε, γρήγορα να προωθούνται στοιχεία ριζοπαστικοποίησης. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε Ε, να έχουμε διαβάσει ένα συγκεκριμένο άρθρο ε, σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και μετά να αρχίζουμε να κατακλυζόμαστε από τέτοιου είδους άρθρα. Επομένως, έρασμος, ε, συμπεριλήψη και ε, παρακολούθηση. Πιστεύω ότι ήδη από τα σχολεία θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, ήδη από τώρα θα επιμείνουμε έτσι ώστε να αναπτυχθούν δράσεις. Και για τα παιδιά που δεν είναι στο σχολείο, όταν ξέρουμε ότι ένα παιδί στα πέντε από μη ευνοημένο περιβάλλον δεν πηγαίνει στο σχολείο, είναι γεγονός ότι ότι ο έρασμος θα πρέπει ε, να υπογραμμίσει και τις μικρές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, αυτές ε, που αφορούν την μη τυπική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φραντς, θέλετε κάποια επερώτηση ή σύντομα σας παρακαλώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είμαστε proactive Ποια είναι η άποψή σας ε, σχετικά ε, με το Ταμείο ε, της Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τα, για παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο γιατί υπάρχει αυτή η αντιρωμά νοοτροπία, όχι επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα τα να μείνουν στο, στο σχολείο. Κοιτάξτε, ο τίτλος μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά εγώ θα ήθελα να πάμε παραπέρα. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περιμένουμε λίγο και με προσοχή να δούμε τι έχουμε και τι θα κάνουμε με το νέο ε, ταμείο. Τι κάναμε ε, με τα χρήματα τα οποία ε, διατέθηκαν ή είναι στη διάθεσή μας με το παρόν ταμείο, γιατί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία δαπανώνται να δίνουν την δυνατότητα να αλλάξουν και κάποιοι κανόνες, να δίνουν την δυνατότητα ε, η συμπερίληψη να γίνει το κεντρικό στοιχείο του προγράμματος και βεβαίως να αφήσουν και χώρο για αυτό που είπα στην αρχή, think out of the box, ρηξικέλευθη διαφορετική σκέψη. Πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε διαφορετικά αποτελέσματα απέναντι σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Γκαμπριέλ. Κυρία Γιώβεβα από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα ή θα σας καλωσορίσω στη δική σας γλώσσα. Στην γραφτές σας απαντήσεις που στείλατε, κυρία υποψήφια Επίτροπε, είπατε ότι θα υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη για καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στο τρίγωνο της γνώσης, όπως οκαλείται έρευνα, καινοτομία, παιδεία και να παρέχετε χρηματοδότηση για τους επιστήμονες, ούτως ώστε να προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μπορείτε να εξηγήσετε πώς θα στηρίξετε τα κράτη-μέλη. Πιο συγκεκριμένα, πώς θα εξασφαλίσετε τη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του τριγώνου της γνώσης με ε, τις αναγκαίες υποδομές από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για το τρίγωνο της γνώσης, έχω υπόψη τον Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογίας, διότι τα ενσαρκώνει αυτά. Όπως είπα, θα ήθελα ε, να ασχοληθώ περισσότερο με τις διάφορες κοινωνίες καινοτομίας και να δω τι έκαναν για τα κράτη-μέλη. Δύο πράγματα βλέπω πολύ συγκεκριμένα που θα κάνουμε αυτά. Όπως σας είπα, και τώρα έχουμε ένα μηχανισμό όπως το Policy Support Facility. Έλαβα υπόψη ότι όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν αυτό το μέσο. Σημαίνει ότι σε όλα τα κράτη-μέλη υπήρξαν αναλύσεις, συστάσεις συγκεκριμένες όταν μιλάμε κυρίως για peer review, εξέταση ομοτήμων, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν αυτά που λέγονται υπόψη στα τρία χρόνια. Αυτό πρέπει να κάνω πρώτα με τα κράτη-μέλη είναι να δω στα πλαίσια του εν λόγω μηχανισμού τι αναλύσεις έγιναν όσον αφορά τα εθνικά συστήματα έρευνα και καινοτομίας, τι συστάσεις έγιναν, τι έγινε και μετά από αυτό μαζί με τα κράτη-μέλη θα συζητήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες που προσφέρονται στα κράτη-μέλη από τον ορίζοντα 2020 και μετά από το ορίζον Ευρώπη και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Για μία ακόμη φορά ερχόμαστε σε αυτό το θέμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα κράτη-μέλη να έχουν ε, σαφή γνώση αυτών που υπάρχουν. Τον, του Ταμείου, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι το Κοινωνικά Ταμεία και το Invest EU, τι δυνατότητες έχουν. Για μένα, εγώ θα έδινα ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα παραδείγματα, συστάσεις που αφορούν συγκεκριμένα μέτρα. Και μετά, μαζί με τα κράτη-μέλη, να δούμε τι δυνατότητες χρηματοδότησης υπάρχουν για να τους δώσουμε αυτό το συνέστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή τις συστάσεις που τους δίνουμε. Και αυτά που διατυπώνουν οι εμπειρογνώμονες είναι συστάσεις που πραγματικά είναι υλοποιήσιμες. Θα εργαστώ επ' αυτού αν έπρεπε να επελέξω, διότι υπάρχουν και άλλες ε, προσεγγίσεις. Εγώ περιγράφω λύσεις όπου μαζί με τα κράτη-μέλη μπορούμε από κοινού να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Διευκρινιστική ερώτηση, ορίστε. Ευχαριστώ. Πώς προτίθεστε να εφαρμόσετε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετάβαση προς μια δίκαιη κοινωνία και μια κοινωνία που θα είναι ουδέτερη όσον αφορά το κλίμα. Απάντηση. Έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Παιδεία, έρευνα και ανατομία πρέπει να τα δούμε μαζί. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό θεωρώ πρόκληση. Γι' αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι πραγματικά μια ευκαιρία. Αρκεί να δείτε το πώς θέλουμε να ζωγονίσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας και ήδη από τώρα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε με την παιδεία. Δεν θα είναι εύκολο. Όταν τα βλέπουμε αυτά και βλέποντα τι εσωτερικέ διεργασίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβανόμεθα ότι μεγάλη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί γι' αυτό. Προφανώ θα φροντίσω ότι στο τέλο να έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική τη γνώση που θα καλύπτει την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία. Αλλά πριν να ονειρευτώ, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να δώσουμε περισσότερο περιεχόμενο σε όλα αυτά. Μετά, όπως είπα, με το πρόγραμμα Horizon 2020 έχουμε δυνατότητες πραγματικά να φροντίσουμε το ώστε η έρευνα να εξυπηρετεί την καινοτομία, καινοτομία να εξυπηρετεί την έρευνα. Έδωσα ήδη παραδείγματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Καινοτομίας, αλλά ήδη αναφέρθηκα και στον επιταχυντή. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που είναι pathfinders, διερευνούν, είναι χνηλατικά ε, λοιπόν, θα πρέπει να στοχεύσουμε την έρευνα για να ανακαλύψουμε τεχνολογία και μετά η τεχνολογία ρηξικέλευθη με τον επιταχυντή θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην αγορά. Ιδού ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση είναι από την Μαρία Τικράσα Καρβάλια, η οποία είναι ε, συντονίστρια από την Ήτρε και από το ΕΛΚΑ. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε και κυρία Υποψήφια Επιτροπέ Μαρία Γκαμπριέλ, σας καλωσορίζω και εγώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την βιομηχανική ηγεσία. Θα κάνω μία δήλωση και στη συνέχεια θα θέσω τις ερωτήσεις μου. Πιστεύω ότι χωρίς επιστήμη η έρευνα σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ δύσκολο να πετύχει τις κλιματικές μας ε, φιλοδοξίες και να εξασφαλίσει μια ισχυρή βάση την οποία θέλουμε να έχουμε ε, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική μας ε, βάση στην Ευρώπη. Μια βιομηχανική στρατηγική λοιπόν θα έχει στον πυρήνα της την επιστήμη και την πολιτική καινοτομία και ένα σύστημα το οποίο θα κάνει τους επενδυτές να επενδύουν σε διάφορους τομείς, στα τρόφιμα, στο, στην αεροπορία, στα χημικά, στις δημιουργικές βιομηχανίες. Έχω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Τι συγκεκριμένες προτάσεις έχετε στην πολιτική σας και στον ορίζοντα Ευρώπη για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ισχυρή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Και πώς πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των βιομηχανίας προκειμένου να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καμπριέλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Όντως, είπαμε ότι η ικανότητα αυτής ε, της Ευρώπης βασίζεται στην βιομηχανία μας. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, πρώτη μα μας αυτή σε βιομηχανικό επίπεδο. Θα πρέπει να επενδύσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα να επενδύσουμε με στρατηγικό σκοπό στρατηγικό τρόπο για να δούμε πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και μια και θέσατε τα θέματα τη βιομηχανία, να διευκρινίσω το εξή αυτή τη εξαρχή ότι πρόκειται για μια συνεργασία που πρέπει να υπάρξει με την ε, πρόεδρο Γκουλάρ και με την αντιπρόεδρο Φεστάγκερ. Γιατί θα πρέπει να θέσουμε το στόχο της νέας βιομηχανικής στρατηγική στην Ευρώπη. Αυτό που θεωρώ ότι είναι ε, σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι χωρίς έρευνα και καινοτομία δεν θα μπορέσουμε ε, ρεαλιστικά να κάνουμε έξυπνες επενδύσεις και να φροντίσουμε η συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα να λεφτεί υπόψη. Σωστά επισημάνατε σε τι βαθμό εξαρτάται η επίτευξη των στόχων για το κλίμα από την κοινοτομία και τι προτεραιότητα αποτελούν. Στον ορίζοντα 2020 ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή και συνεχίζεται στον ορίζοντα Ευρώπη. Επισέρχονται λοιπόν στοιχεία καινοτόμα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, ψηφιοποίηση, αλλαγή του κλίματος, βιομηχανοποίηση, Όλα αυτά λοιπόν τα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και των προγραμμάτων flagship, των προγραμμάτων ορόσημα, γιατί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις που έχουμε κάνει. Θα δείξω μεγάλη προσοχή λοιπόν προκειμένου στην επόμενη βιομηχανική στρατηγική μέσω της έρευνας και της καινοτομίας η Ευρώπη να επενδύσει έξυπνα, να υποστηρίξει τα ισχυρά της σημεία και να μην διστάσει να ηγηθεί του επόμενου κύματος εντομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία διευκρινιστική ερώτηση από την κυρία Καρβάλιο. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θα υποστηρίξουμε ένα ανοιχτό και φιλόδοξο πρόγραμμα ορίζοντας Ευρώπης. Ωστόσο, κάτι που δεν έχουμε πετύχει ακόμα στον ορίζοντα 2020 και θέλουμε να το περιλτιώσουμε στον ορίζοντα Ευρώπη. Πείτε μας λοιπόν πώς το κρίνετε αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε καλύτερα το θέμα των ορίων της έρευνας στον ορίζοντα Ευρώπη. Θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιούνται πιο καλά σε συγκεκριμένε εφαρμογέ, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά συνεργασίε ιδιωτικού και α, δημοσίου κλάδου. Αναφερθήκατε στο υδρογόνο, στο Clean Skies. Πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη συνέργεια μετά του ERC και των υπόλοιπων προγραμμάτων και να εφαρμοστούν καλύτερα και τα υπόλοιπα σκέλη του ορίζοντα Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαμπριέλ. Μάλιστα. Πολύ σωστά υπογραμμίζετε αυτήν την ε, πρόκληση. Κοιτάξτε, έχουμε τον πρώτο πυλώνα που αφιερώνεται ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Αριστεία και έχουμε εδώ και τις δράσεις Μαρή Κυρί, Γιατί δεν μπορούμε ε, να τα δούμε αυτά και στις διάφορες αποστολές του πυλώνα 2, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε επίσης και στα πλαίσια των εργασιών που ε, ο ΠΟΕ έχει αρχίσει να ε, προωθεί. Ποια είναι τα οικοσυστήματα των ερευνητών. Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να συμβάλλουμε στην έρευνα και όταν βλέπει κανείς τις αποστολές ε, ε, ε, έχουμε επιστήμονες ε, οι οποίοι και για ψηφιακά αγωνίζονται και για το, την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση του καρκίνου. Επομένως μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα των ε, επιστημόνων, των ερευνητών έτσι ώστε και αυτοί να γίνουν περισσότερο proactive. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν ε, να έχει και μία ανακοίνωση στο δεύτερο εξάμεινο του 20 ε, για τον Ευρωπαϊκό Χώρο ε, Έρευνας ε, και εδώ ήδη να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έχουμε εντωμεταξύ προωθήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαλεάν, ολοκληρώθηκε λοιπόν ο χρόνος των ερωτήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τις απόψεις που εκφράστηκαν. Κοιτάξτε, ζητώ συγγνώμη ε, κύριε υποψήφια επίτροπε γιατί αναγκάστηκα να σας διακόψω σε ορισμένες από τις απαντήσεις σας. Θα έχετε όμως τη δυνατότητα να κάνετε μια τελική δήλωση ε, πέντε λεπτών έτσι ώστε να εκφράσετε κάποιες ιδέες τις οποίες ενδεχομένως δεν στάθηκε δυνατόν ε, να εκφράσετε. Σας δίνω λοιπόν τώρα τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που μου έδωσε τη δυνατότητα να πάρω το σφιγμό των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών και να σας διαβεβαιώσω ότι εάν δώσετε το πράσινο φως για τον διορισμό μου ε, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη πορεία ε, ανοιχτού διαλόγου και ε, ειλικρίνειας. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν και ξανακούστηκαν. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι ε, ο τίτλος αφορά και την ε, νεολαία και τον αθλητισμό και την έρευνα και την καινοτομία και την ε, εκπαίδευση. Το widening, αυτή η διεύρυνση είναι πάρα πολύ σημαντική, οι εταιρικέ σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και όπως είπα και προηγουμένως, το ξαναλέω και το υπογραμμίζω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο για χάσιμο. οπωσδήποτε εγώ θα κινηθώ βάσει των δεσμεύσεων που ανέλαβα ενώπιόν σα. Τώρα θα ήθελα ε, να πω το εξής ακόμα μια φορά. Ήρθε η ώρα να ε, ε, κάνουμε λίγο πίσω, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε καλύτερα και να καταλήξουμε σε επενδύσεις οι οποίες θα είναι πιο στοχευμένες και οι οποίες καλύτερα θα ανταποκρίνονται σε αυτήν την ευρωπαϊκή απάντηση που πρέπει να δώσουμε στις παρούσες προκλήσεις. Θα ήθελα επίσης να ε, αναφερθώ σε εκείνες και εκείνους που μετά από την εισαγωγική μου ε, ε, παρέμβαση αναρωτήθηκαν εάν με τη σειρά που ανέφερα τα στοιχεία θα ιεραρχήσω και τις προτεραιότητές μου. Όχι η ε, δημιουργική βιομηχανία, οι νέοι, η ποιοτική εκπαίδευση, οι περιφέρειες, ε, ο αθλητισμός, οι μικρές γλώσσες, ε, ο, πλούσιος πολιτιστικός χαρακτήρας της Ευρώπης οπωσδήποτε θα βρουν τη θέση τους και επομένως αλληλεγγύη, συνεργασία και ανταγωνιστικότητα σαν ε, αντίθετο τρίπτυχο από αυτό που είχε αναφέρει ο Ζακ Ντελόρ. Θα ολοκληρώσω ε, στην Βουλγαρική. Θα ήθελα ε, να σας πω ότι υπάρχει κάτι που μου είναι ιδιαίτερος ε, προσφυλές. Είναι ο βουλγαρικός ε, ύμνος ε, για, την, για τον πολιτισμό. Είναι πραγματικά τα λόγια τα οποία αναφέρονται και στον Μεθόδιο και τον Κύριλο. Μιλάμε για έναν ύμνο ο οποίος έχει έχει δημιουργηθεί πολλά χρόνια πριν. Ένας από τους μαθητές ε, ενός ε, μεγάλου ε, δασκάλου του Στογιάννοφ είχε εμπνευστεί από ένα ποίημα του δασκάλου και μερικά χρόνια μετά δημιούργησε αυτόν τον ύμνο επιστήμης ε, γνώσης ε, που πεανίζεται στα σχολεία. Και λέει ας πάμε προς ένα πιο λαμπρό μέλος, μέλλον συγγνώμη, με γνώση. Ε, ας προχωρήσουμε ε, με την επιστήμη που ε, αγγίζει τις ψυχές μας και που αποτελεί πραγματικά μια, ένα ηλιόλουστο περιβάλλον. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με τον πολιτισμό. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Γκάμπριελ, ευχαριστώ και τις δύο παρούσες επιτροπές. Άκρος ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Μαραθώνιος, ολάκερος. Χρειάστηκε πολύ χρόνο. Υπήρξαμε αποτελεσματικότατοι. Ζωντανή η συζήτηση, καλύφθηκαν πολλές ιδέες. Καλύψαμε όλα τα χαρτοφυλάκια Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ κύριε Χάν για την πολλή συνεργασία που υπήρχε μεταξύ ΚΟΛΤ ε, και Ήτρε για τη οργάνωση της ακρόσης και δίνω το λόγο σε εσάς, κυρία Βερχάιεν. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου κυρία Βερχάιεν δεν την ακούμε. Ε, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαλέν. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω 100% να ευχαριστήσω τα μέλη και των δύο επιτροπών για τις ερωτήσεις που κάνανε και για την υποψήφια επίσης επιτροπό ε, την κυρία Κάμπριελ για τις εκτενέστατες ε, απαντήσεις της. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση όπως και αναμένονταν για ένα τόσο ευρύ χαρτοφυλάκιο το οποίο μας αφορά ιδιαίτερος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Βάλεαν και την γραμματεία ε, της Ήτρε και τους, τη γραμματεία τη Επιτροπή Πολιτισμού για την πολύ καλή συνεργασία και την καλή υποστήριξη. Όπω γνωρίζετε, καθήκον μα επόμενο είναι από κοινού να αξιολογήσουμε αυτά που ακούσαμε σήμερα. Αυτή η αξιολόγηση θα λάβει χώρα 3η, 1η Οκτωβρίου στις 9 σε μια κοινή συνεδρία συντονιστών στο ESP ε, 1G3. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 9 επαναλαμβάνω ESP 1G3 θα συναντηθούν οι συντονιστές και των δύο επιτροπών για να κάνουν την κοινή διαδικασία αξιολόγησης της ακρόασης και για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εκ νέου και τη Μαρία Γκάμπριελ και ανυπομονώ να κάνουμε την αξιολόγησή μας αύριο. Ευχαριστώ πολύ.